Proszę będziemy powoli zaczynać, bo spotkanie Κυρίες και κύριοι, να σας καλωσορίσω. Σήμερα έχουμε μια έκτακτη συνεδρίαση και εξαιρετική. Εξαιρετική διότι ασχολούμαστε με ένα πολύ σημαντικό θέμα, καταρχάς, και εξαιρετική διότι υποδεχόμαστε δύο αξιότιμους προσκεκλημένους. Πριν περάσω στο βασικό ζήτημα της συνεδρίασής μας, θα ήθελα να σας μιλήσω για τα τυπικά. Έχετε λάβει την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε παρατηρήσεις, μπορούμε να την εγκρίνουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν υπάρχει γερμανική διαρημηνία. Ε, ρυθμίστηκε το ζήτημα. Καλώς. Ως προς τη διερμηνία λοιπόν, δεν έχουμε διερμηνία σε ορισμένες γλώσσες, δηλαδή στα μαλτέζικα, στα σλοβακικά και στα εσθονικά μεταξύ άλλων. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω όλους και όλες σας. Θα ασχοληθούμε με τον ανταγωνισμό και την γεωργία. Ο ανταγωνισμός δεν είναι κάτι στο οποίο ε, συχνά μπαίνει σε βάθος η Επιτροπή μας. Συχνά γίνεται λόγος για το ζήτημα του ανταγωνισμού, πάντοτε όμως χρησιμοποιούμε γενικούς όρους και δεν έχουμε συχνά χρόνο να αναλύσουμε σε βάθος το θέμα του ανταγωνισμού στη Γεωργία, να αναλύσουμε σε βάθος τον ανταγωνισμό ε, σε όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Ενώ είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό και για την εσωτερική και την εξωτερική αγορά της Ένωσης. Πρέπει να έχουμε σωστή μορφή ανταγωνισμού, καλές εμπορικές πρακτικές, γιατί όλα αυτά επηρεάζουν την τύχη των αγροτών. Επηρεάζουν τα εισοδήματα που μπορούν να αποκομίσουν από τη δραστηριότητά τους. Θα ήθελα θερμά να ευχαριστήσω τους δύο προσκεκλημένους μας. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που σας υποδέχομαι εδώ σήμερα. Να καλωσορίσω την Επίτροπο Μάργαρετ Φεστάγκερ Βεβαίως και χαίρομαι διότι είναι παρόν μαζί μας ο Επίτροπος κύριος Σχόγκαν. Όμως τον κύριο Χόγκαν τον βλέπουμε πιο συχνά συνεργαζόμαστε πιο συχνά και χαίρομαι ιδιαίτερως που σας καναβλέπω κύριε Χόγκαν εδώ. Το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής να αναλύσει σε περισσότερο βάθος τα ζητήματα του ανταγωνισμού. Θέλουμε την ε, εσωτερική και εξωτερική άποψη για το θέμα αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει τις εργασίες μας για το θέμα του ανταγωνισμού και πώς επηρεάζει ορισμένες αρρώσιμες καλλιέργειες ή πώς επηρεάζει την παραγωγή βόηου κρέατος. Έχουμε έγραπτα συμπεράσματα και σήμερα λοιπόν θα ακούσουμε τις απόψεις των ομιλητών μας. Έχουμε μια μισή ώρα συζήτηση. Στις 8.30 θα ξεκινήσει η ψηφοφορία. Δεν βλέπω τον κύριο Νίκολσον στην αίθουσα. Ελπίζω ότι θα είναι στην ώρα του. Μάλλον ε, δουλεύει τις τροπολογίες μέχρι η τελευταία στιγμή. Πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες έχουν κατατεθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά αργότερα. Και να δώσω το λόγο στους επιτρόπους. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο θέλει να μιλήσει πρώτος. Καλώς ορίσατε. Παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή που προσκάλεσε την Επίτροπο Φεστάγκερ και μένα να συζητήσουμε το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τις κοινέ πωλήσει από αγρότες σε τρεις βασικούς τομείς της γεωργίας. Και με χαρά έχουμε αυτή την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις με εσά σήμερα για το θέμα αυτό. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν έχουν κοινού στόχου στον τομέα τη γεωργία. Θέλουμε ο, γεωργικό τομέα να είναι πιο ισότιμο και πιο ανταγωνιστικό. Αυτά μα είπατε ε, στην, ε, στις προτάσεις για τη μεταρρύθμιση. Θέλουμε ο αγροτικός τομέας να είναι πιο πράσινος και πιο βιώσιμος, πιο αηφόρος. Έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη, τις κατευθυντήρης γραμμές, αλλά ας δούμε το ιστορικό υπόβαθρο. Καταρχάς, για να δούμε την ευρύτερη εικόνα. Ο ανταγωνισμός είναι καθημερινότητα, καθημερινή πραγματικότητα για πολλούς ε, παραγωγούς γεωργικών ε, προϊόντων στις περισσότερες αγωγές, α, αγορές και αυτό είναι λογικό. Μετά από διάφορες μεταρρυθμίσεις στην κοινή γεωργική πολιτική η δική μας πολιτική γεωργική βασίζεται περισσότερο από ποτέ στην αγορά. Οι αγρότες μας αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικές προκλήσεις, αλλά και οι καταναλωτές αυξάνουν τις απαιτήσει τους που θέλουν καλύτερα προϊόντα, αηφόρα βιώσιμα προϊόντα, ε, ανιχνεύσιμα προϊόντα. Και οι αγρότες αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από τις μη ευρωπαϊκές εισαγωγές. Έχουν εμπορικούς εταίρους πολύ ισχυρούς. Τους, όσους κάνουν την επεξεργασία, τους επιχειρήσεις λιανικής, δεν έχουν μεγάλη διαπραγματευτική ισχύ οι αγρότες έναντι των μεγάλων αγοραστών. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τους αγρότες να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις. Ο νομοθέτης με την παράδο των ετών έχει σχεδιάσει ένα σύνολο κανόνων για έναν ευρωπαϊκό γεωργικό τομέα που θα είναι πιο ισότιμος, πιο πράσινος, πιο ανταγωνιστικός, πιο αηφόρος. το Κοινοβούλιο και η δική σας Επιτροπή διαδραματίζει ένα καθοριστικό ρόλο ως προς αυτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι η πολιτική ανταγωνισμού και η πολιτική γεωργίας έχουν μια ειδική σχέση. Βάσει των κανόνων ανταγωνισμού, πρακτικές όπως οι ομαδικές πωλήσει προϊόντων αποτελούν περιορισμό του ανταγωνισμού και απαγορεύονται, εκτός και αν αποδειχθεί ότι ευνοούν τους καταναλωτές. Όμως στη Γεωργία αυτό είναι διαφορετικό. Υπάρχουν εξαιρέσεις για συμφωνίες και επιχειρηματικές πρακτικές που επιδιώκουν και βοηθούν την επίτευξη των στόχων της κοινή γεωργικής πολιτικής. Γι' αυτό ο νομοθέτης, δηλαδή εσείς και το Συμβούλιο, έχει αποφασίσει ότι οι βασικοί κανόνες ανταγωνισμού θα ισχύουν στο γεωργικό τομέα, αλλά θα υπόκεινται σε έναν αριθμό εξαιρέσεων. Με νομικό λεξιλόγιο εδώ μιλούμε για, ε, χρησιμοποιούμε τον όρο ε, παρεκκλήσεις. Τα, εδώ και 50 χρόνια ισχύει η κοινή γεωργική πολιτική και ο νομοθέτης έχει οθετήσει διάφορες ε, παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις μπορούν οι αγρότες στην Ευρώπη να δράσουν από κοινού στην αγορά και με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής και υπέβαλε προτάσεις για νέες εξαιρεσει από τον ανταγωνισμό. Προσθέσατε νέους κανόνες στις αρρώσιμες ή αρωτρέες καλλιέργειες, στο βόιο και μοσχαρίσιο κρέας και στο ελαιόλαδο. Οι νέοι αυτοί οι κανόνες ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα αιτήματα των παραγωγών ε, που θέλουν τα μέτρα να ενισχύουν τη διαπραγματευτική τους ισχύ έναντι των αγοραστών τους. Όταν λοιπόν ε, ασχολείται με αυτά τα αιτήματα ο νομοθέτης υιοθετεί ισορροπημένη προσέγγιση. Θέλει ο νομοθέτης ε, οι αγρότες να συνεργαστούν περισσότερο, να ενσωματώσουν τις δραστηριότητες τους για να έχουν ένα κοινό εγχείρημα αποτελεσματικό και αηφόρο. Θα μπορούσαν να έχουν μια κοινή ε, πλατφόρμα διανομής για περισσότερη ευελιξία, αξιοπιστία και ταχύτητα στη διανομή. Εάν οι αγρότες δουλέψουν μαζί, συνεργαστούν με αυτόν τον τρόπο, τότε έχουν πολλές πιθανότητες να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και μπορούν μάλιστα να αντιμετωπίσουν τους αγοραστές και τα υπόλοιπα μέλη της ε, εμπορικής αλυσίδας που ασχολούνται με τη την επεξεργασία, τη συσκευασία, τη, τη λιανική πώληση και μπορούν να ε, αντιπαρέλθουν εμπορικές πρακτικές που οι αγοραστές ε, τυχόν τους επιβάλλουν. Η προσέγγιση αυτών των νέων εξαιρέσεων μας βοηθάει να πετύχουμε τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής στους τρεις αυτούς κλάδους, τομείς της γεωργίας. Έτσι έχουμε καλύτερα εισοδήματα για τους αγρότες, αυξημένη παραγωγικότητα, περισσότερη διαθεσιμότητα των τροφίμων, των προμηθειών και λογικές τιμές για τον καταναλωτή. Άλλωστε γι' αυτό προσπαθούμε να έχουμε γεωργικό τομέα που να είναι ανταγωνιστικός και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του ανταγωνισμού και εντός και εκτός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι νέοι κανόνες ε, αυτοί περιλαμβάνονται σε άρθρα 169-171 του κανονισμού για την κοινή οργάνωση της αγοράς. Καθίσταται σαφές ότι οι αγρότες σε αυτού του τομεί μπορούν να έχουν ομαδικέ πωλήσει και να καθορίζουν τιμέ, όγκου παραγωγή και άλλου όρου στην εμπορική συναλλαγή και μπορούν να το κάνουν εάν ε, οι όγκοι που, ε, τα μεγέθη δηλαδή που εμπλέκονται εκεί είναι λογικά. 15% για το βόλιο και μοσχαρίσιο κρέα, 20% για το ελαιόλαδο. Και αν έχουν βεβαίω οργανωθεί σε μια οργάνωση παραγωγών ε, που διενεργεί και άλλε δραστηριότητε. Μπορεί να έχουν κοινή διανομή, κοινή αποθήκευση, να είναι πιο αποτελεσματική με αυτόν τον τρόπο. Για να πετύχουμε λοιπόν τους στόχους της κοινή γεωργικής πολιτικής χρειάζεται σωστό σημείο ισορροπίας, να έχουν περισσότερη διαπραγματευτική ισχύ οι αγρότες και να μην υπάρχουν μονοπόλια, δομές μονοπωλιακέ. Αυτά ως γενικό ιστορικό υπόβαρο θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο Φεστάγκερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Φυσικά Συμφωνώ απολύτως με τον συνάδελφό μου. Να πω όμω λίγα λόγια για τη δουλειά μας μέχρι τώρα. Δεν αρκεί να έχουμε κανόνες. Θα πρέπει να εφαρμόζονται, θα πρέπει να γίνουν η, ε, πραγματική, η πραγματικότητα και η καθημερινότητα για τους αγρότες και για τους ε, χρήστες των ε, κανόνων αυτών. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι, κατανοητοί και να δίνουν πραγματικές κατευθυντήριες γραμμές, διότι αλλιώς πάει χαμένη όλη η δουλειά που κάνετε εσείς ως νομοθέτες. Η Επιτροπή σας μας κάλεσε να φροντίσουμε να υπάρχει περισσότερη συνέπεια όσον αφορά την εφαρμογή του νόμου σε όλα τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε και αυτό είναι ο λόγος που η Κομισιόν εξέδωσε ε, το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών που συζητάμε σήμερα. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Οι αποκλήσεις μεταξύ κρατών μελών ε, δεν προσφέρουν συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Οι κατευθυντήρες γραμμές αποτελούν κοινή προσπάθεια της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας. Έχουμε καλέσει όλους να του, τις σχολιάσουν, γεωργούς και αρχές και φυσικά την Επιτροπή σας. Ο λόγος που καλέσαμε όσο γίνεται περισσότερους να σχολιάσουν το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών είναι για να διασφαλίσουμε την χρησιμότητά τους. Όχι πως δεν είναι χρήσιμες όλες οι κατευθυντήριες, γραμμέ κατευθυντήριες γραμμές της Κομισιόν, αλλά χρήσιμο είναι, σημαντικό είναι να μπορούν να εφαρμοστούν άμεσα, να μην χρειάζεται κάποια μετατροπή. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι οι νέοι ότι οι γεωργοί θα πρέπει να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς. Θα πρέπει οι ίδιοι να αξιολογήσουν την συμμόρφωσή τους με τους κανόνες. Για να το κάνουν αυτό χρειάζονται κατανοητές κατευθυντήριες γραμμές. Διότι αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να αποτελούν εγχειρίδιο για να γίνει αυτή η δουλειά και θα πρέπει να δίνουν παραδείγματα σχετικά με την ε, εφαρμογή των κανόνων σε διάφορες ε, καταστάσεις. Διάφοροι συμμετέχοντες ε, στη δημόσια διαβούλευση τόνισαν τη χρησιμότητα και ζήτησαν περισσότερα πρακτικά παραδείγματα. Οι υπηρεσίες μας ασχολούνται τώρα με αυτό ώστε να γίνουν πιο χρήσιμες οι κατευθυντήρε γραμμές και από αυτήν την άποψη. Θέλουμε να είναι φιλικές προς το χρήστη και να επιτρέπουν στους γεωργούς και στους παραγωγούς να εφαρμόζουν ε, εύκολα και ομαλά τις κατευθυντήρε αυτές γραμμές. Σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι οι κατευθυντήρε γραμμές ε, δεν ε, επιβάλλουν νέε διαδικασίε, νέε προϋποθέσεις και νέες απαιτήσεις. Η Κομισιόν περιορίστηκε στην ε, ερμηνεία, στην επεξήγηση των νέων κανόνων που υιοθέτησε ο νομοθέτης. Είναι σημαντικό το ότι αυτές οι κατευθυντήρες γραμμές αποτελούν αποτέλεσμα μιας εντελεχούς διαβούλευσης των εθνικών ε, αρχών ανταγωνισμού και των Υπουργείων Γεωργίας ακόμα πριν γίνει η δημόσια διαβούλευση. Η διαβούλευση αυτή στόχο είχε να διασφαλίσει οι κατευθυντήρες γραμμές να αντικατοπτρίζουν ε, τις ε, διάφορες πτυχές των τομέων αυτών. Όπως μόλις τόνισε ο Επίτροπος Χόγκαν, αρκετοί κανόνες που ισχύουν για άλλους τομείς δεν ισχύουν για τον ε, τομέα της γεωργίας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε στενά με τις εθνικές αρχές, τους γεωργούς και τα Υπουργεία, ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, Ελπίζουμε ότι οι κατευθυντές αυτές γραμμές θα επιτρέψουν κοινή και ενιαία εφαρμογή των νέων κανόνων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών ήταν αντικείμενο πολύ χρήσιμων ε, παρατηρήσεων κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης και όπως γνωρίζετε λάβαμε και σημαντικές παρατηρήσεις από την Επιτροπή σας. Είμαστε ευγνώμονες που καταβάλατε την προσπάθεια αυτή και η γραπτή σας συνεισφορά όπως και τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης θα ληφθούν υπόψη κατά την τελική επεξεργασία των κατευθυντηριών γραμμών. Επιτρέψτε μου να σχολιάσω ένα ή δύο πράγματα. Ζητήσατε τις απόψεις μας σχετικά με τις γενικές αποκλίσεις ε, όσον αφορά τις επιχειρηματικές πρακτικές ε, στον γεωργικό τομέα. Αυτά προβλέπονται στο άρθρο 206 έως 209 της κοινή οργάνωσης αγοράς. Ο Επίτροπος Χόγκαν και εγώ επικεντρωθήκαμε στις ε, νέες διατάξεις του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι οι κατευθυντήρες γραμμές καλύπτουν την κοινή πώληση από τους παραγωγούς στους τομείς ε, ελαιολάδου, βοήου κρέατος ε, και αρωτρέων ε, καλλιεργιών. Οι κανόνες αυτοί είναι καινούριοι. Οι παραγωγοί στους τομείς αυτούς χρειάζονται περαιτέρω διευκρινήσεις σχετικά με τους κανόνες στους τομείς αυτούς. Όσον αφορά άλλους γεωργικούς τομείς, οι υπηρεσίες της Κομισιόν ζήτησαν προσανατολισμό από έναν τομέα, τον τομέα της ε, ζάχαρης. Αυτό είναι λογικό καθότι η παραγωγή ζάχαρης θα αντιμετωπίσουν νέες συνθήκες από το 2017, ε, από το 2017 και μετά λόγω σημαντικών αλλαγών που έχουν γίνει όσον αφορά το ε, νομικό καθεστώς. Τώρα εξετάζουμε εάν χρειαστεί περαιτέρω προσανατολισμός. Επίσης αναφέρατε την ανάγκη για περισσότερες οδηγίες όσον αφορά τον ορισμό των ε, αγορών και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης ε, στην αγορά. Υπάρχουν ε, κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον ανταγωνισμό που μπορούν να δοθούν σε παραγωγούς και άλλους ενδιαφερομένους για να μπορούν ε, να τι εφαρμόσουν. Οι υπηρεσίες μας ε, είναι στη διάθεση ε, των ενδιαφερομένων για να παράσχει περαιτέρω βοήθεια και πληροφόρηση. Κλείνοντας, να πω λίγα λόγια σχετικά με το πού βρισκόμαστε στην όλη διαδικασία εξετάζουμε τις παρατηρήσεις που λάβαμε στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε στις 15 Μαΐου. Θα οριστικοποιήσουμε την επεξεργασία με βάση τις παρατηρήσεις που θα ακούσουν απόψε. Συμφωνήσαμε με την Επιτροπή σας να μπορείτε να εκφράσετε τη γνώμη σας ε, πριν τα τελικά βήματα και ακριβώς γι' αυτό πραγματοποιείται η σημερινή συνεδρίαση. Αποτελεί το τελευταίο βήμα προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητήσει την άποψη των συμβουλευτικών, της Συμβουλευτικής Επιτροπής ε, των ε, Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού και η Επιτροπή αυτή θα συγκληθεί τον Σεπτέμβριο. Μετά θα υποβάλουμε τις κατευθυντήρες γραμμές στο Σώμα των Επιτρόπων για να υιοθετηθούν. Αυτό θέλουμε να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα το ε, φθινόπωρο. Και ο Επίτροπος Χόγκαν και εγώ παραμένουμε αφοσιωμένοι στην δουλειά αυτή, διότι οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τον ανταγωνισμό. Γι' αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να λειτουργήσουν σωστά οι κατευθυντές γράμμες αυτές, να είναι συγκεκριμένες και κατανοητές. Νομίζω ότι και οι γραπτές παρατηρήσεις της Επιτροπής σας αλλά και η σημερινή συνεδρίαση θα μας επιτρέψουν να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Apeluję też, abyśmy korzystali z tej formy pisemnej komentarzy, o Προτείνω να χρησιμοποιήσουμε, όπως προτείνει η κυρία Επίτροπο στην γραπτή διαδικασία. θα ξεκινήσουμε με παρεμβάσεις των συντονιστών. Θα ήθελα να δηλώσετε όλοι πόσοι, ποιοι θέλετε να μιλήσετε για να οργανώσουμε λίγο το χρόνο ομιλίας. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μέχρι τις 8.30. Ε, οι συντονιστές ε, θα μιλήσουν πρώτα, δεν έχουν, ε, δεν έχουν όριο χρόνο, αλλά να είναι σύντομοι αν γίνεται παρακαλώ. Και ως δες πρώτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ Χιόγκαν, βέστα Βέσταγκερ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε παρόντες. Δεν θα μιλήσω μέχρι τις 8.30. Ε, αν και θα, ήταν, ε, αν και θα ήμουν ικανός να κάνω κάτι τέτοιο. Σας ευχαριστώ πολύ που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα σήμερα. Είναι θέμα που αφορά όλους μας ε, και εντός του ΕΛΚ συζητάμε συχνά το θέμα αυτό. Η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχω εδώ το κομπέντιουμ σχετικά με την ε, μεταρρύθμιση ε, την αγροτική στα κράτη-μέλη και από ό,τι βλέπω έχουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που δεν είχαμε πριν 10 ε, χρόνια. Αυτό όμως συνάδει με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι ο συνάδελφος Νταντάν μπορεί να λαμβάνει συνδεδεμένε πληρωμέ, ενώ στη Γερμανία δεν, το, δεν γίνεται αυτό. Τότε μήπω θα πρέπει και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση σχετικά με τι συνδεδεμένε πληρωμέ ε, και έτσι θα υπάρξει μεγάλη πίεση ε, στην Ευρώπη. για να έχουμε ίσες ε, συνθήκες ανταγωνισμού. Για παράδειγμα στο βόλιο Κρέας. Εν πάση έχουν ληφθεί αποφάσεις ε, και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε, τις σημαντικότερες ε, στρεβλώσεις ανταγωνισμού τις έχουμε ε, σε τομείς όπου η Ευρώπη δεν έχει αρμοδιότητες. Ε, για παράδειγμα, στην φορολογία. Στη Δανία δεν φορολογείται το ντίζλ για γεωργική χρήση. Σε άλλες χώρες όμως ναι, αυτό είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η φορολογική νομοθεσία όμως είναι εθνική αρμοδιότητα. Οι Δανία αντιθέτως πρέπει να πληρώσουν ε, υψηλά τέλη για την ε, χρήση φυτοφαρμάκων. Έχουμε περιβαλλοντικά τέλη που επίσης ενδιαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, αλλά και αυτό αποτελεί εθνική αρμοδιότητα και ο πρόεδρος Γιούγκερ πρότεινε τα κράτη-μέλη να μπορούν μόνα τους να αποφασίσουν όσον αφορά την εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να αποτρέψουμε την Επιτροπή από το να υιοθετήσει τέτοια απόφαση. Επίσης, όσον αφορά τις ε, τιμές ε, στην ε, Ευρώπη ε, σχετικά με την αναπαυσία. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες διαφορές ή τις τιμές της ενέργειας που επίσης αποτελούν εθνική αρμοδιότητα. Στο biodiesel ίσως θα μπορούσε η Ευρώπη να βρει μια ρύθμιση ώστε να χρησιμοποιείται αυτό το καύσιμο. Ε, περιμένω με αγωνία να δω τις ε, κατευθυντήριες γραμμές και ελπίζω να ε, έχουν καλό αποτέλεσμα. Μιλάμε για ενίσχυση του παραγωγού. Εδώ και πολλά χρόνια είμαι πρόεδρος σε, μια συνομοσπονδία που παράγει, σε ένα συνεταιρισμό που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα. Είχαμε λοιπόν ένα προϊόν ε, με έναν παραγωγό στο νότο της, Ευρώπη, της Γερμανίας και έναν ε, στη, στο βορρά. Η διαμόρφωση των τιμών ε, είχε γίνει πολύ καλά, αλλά κατόπιν είδαμε έναν μικρό παραγωγό από άλλο κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατέστρεψε όλη τη διαμόρφωση των τιμών. Ένας μικρός παραγωγός δηλαδή ανέτρεψε όλη την κατάσταση. Φαντάζομαι ότι και οι συνάδελφοι θα έχουν να κάνουν παρατηρήσεις. Δεν θέλω λοιπόν ε, να ε, μιλήσω πολύ χρόνο. Αλλά ε, αναφέρθηκε ο τομέας της ζάχαρης, έχουμε και τον τομέα του γάλακτος. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και περιμένω με αγωνία να δω τις κατευθυντές γραμμές. Ευχαριστώ. Κύριος Δεκάστρο, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα, προσπαθώ, θα προσπαθήσω εγώ να βουτήξω κάποια λεπτά από το συνάδελφο Ντές. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Βεστάγκερ και τον κύριο Χόγκαν για την παρουσία τους εδώ. Είναι ενδιαφέρον να δούμε το θέμα του ανταγωνισμού και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού σε έναν ε, τομέα όπως αυτό της γεωργίας που όπως ε, είπε ο συνάδελφος Ντες ε, θα είχε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αυτό που σήμερα ωστόσο είναι σημαντικό είναι να συμβάλλουμε ως Επιτροπή στο θέμα των παρεκκλήσεων που συζητήσαμε και που η ανακοίνωσή σας μέσω των καθοδητήριων γραμμών προσπαθεί να αντιμετωπίσει ιδίω τους τρεις τομείς, ελαιόλαδο, ε, σπόδι προσφορά και ε, βόλιο. Εγώ θα κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις που ισχύουν για όλο τον τομέα. Η γεωργία είναι ένας ε, ιδιαίτερος κλάδος οικονομικά χαρακτηρίζεται ως price taker, δεν μπορεί να επηρεάσει σχεδόν καθόλου την τιμή σε σχέση με τους κλάδους που είναι παραπέρα όπως η βιομηχανία ε, και που έχουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα συγκέντρωσης από τη γεωργή. Το πρόβλημα λοιπόν γεννάται από την ικανότητα της πολιτικής να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στην συνένωση, συνένωση των γεωργών προθώντας ισχυρότερες οργανώσεις γεωργών για να αντισταθμίσουν του κατόπιν βρίσκουν, πριν ή μετά βρίσκουν οι γεωργοί ε, απέναντί τους. Άρα αυτές οι καθοητήρες γραμμές είναι που θα πρέπει να δώσουν τις δυνατότητες στους γεωργούς μέσω των αυτοδηλώσεων τους να μπορέσουν με καλύτερο τρόπο και με μεγαλύτερη προσοχή να χρησιμοποιήσουν τις παρεκκλήσεις που εισάγαμε και που χάρη στον ε, συνάδελφο για το ενιαίο πρόγραμμα στην περασμένη θητεία μπορούμε να διευρύνουμε. Διευκρινίζοντας σαφώς λοιπόν πώς ε, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία αυτά από πλευράς γεωργών που συχνά δεν το ξέρουν και σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι υπάρχει μεν το εργαλείο αλλά εφαρμόζεται λίγο παρά μόνο σε ακραίες ε, ανάγκες ε, που πρέπει να μας δείξει ακριβώς την ανάγκη καλύτερης συγκέντρωσης και οργάνωσης των γεωργών για να αντιμετωπίσουν την συγκέντρωση που υπάρχει στους προγενέστερους και μεταγενέστερους τομείς της δραστηριότητας αυτής. Εγώ να ευχαριστήσω λοιπόν. Το θέμα της στρέβλωσης του ανταγωνισμού είναι τεράστιο, αλλά στον τομέα αυτό νομίζω ότι η δουλειά που κάνετε είναι πολύ σημαντική. Θα προσπαθήσουμε να το εξηγήσουμε κάπως καλύτερα και στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Συχνά οι αρχές ανταγωνισμού οι δομές αντιτράστ δεν αντιλαμβάνονται την διαφορετικότητα της γεωργίας σε σχέση με, τους, με τους υπόλοιπους κλάδους. Εμείς έχουμε έναν ε, γεωργικό τομέα που, που, υποφέρει από τις χαμηλές τιμές για παράδειγμα, αλλά στην πράξη άλλοι τομείς ε, πιο πέρα από τη γεωργία εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση ενώ στην ουσία η γεωργία μόνο την υφίστανται ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Επίτροπε Χόγκαν, επίτροπε Βεσάγκια Χέρ, είναι θετικό ότι ενισχύεται τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τον αγωνισμό οι γεωργοί. Πολλοί γεωργοί αισθάνονται συμπιεσμένοι μεταξύ άλλων πλευρών της αλυσίδας ε, διατροφής. Φερρυπίν, στη προγενέστερα ε, λιπάσματα, μηχανήματα και μεταγενέστερα ο κλάδος της μεταποίησης. Ε, κάποιες πρωτοβουλίες, αυτέ ε, αυτές όντως δείχνουν τα προβλήματα. Θα έπρεπε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στις ζωέ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Ζητώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, κύριε Επίτροπε τι μπορείτε να κάνετε ως αρμόδια τον ανταγωνισμό για να παρακολουθείτε συνεχώς την κατάσταση των εισρωών στη Γεωργία και να παρεμβαίνετε όταν υπάρχουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Σενέρα. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Μπήκα τώρα μόλις, λυπάμαι που δεν μπόρεσα να είμαι νωρίτερα εδώ και δεν άκουσα τι μας είπαν. Πάντως, θέλω να κάνω κάποιες σκέψεις για το θέμα του ανταγωνισμού μας έλεγαν ότι οι κανόνες ανταγωνισμού ήταν περιτές για την προστασία των καταναλωτών, ήταν αναγκαίες για να προστατεύσουν τον καταναλωτή και να υπάρχουν ισορροπημένες τιμές. Ωστόσο, αυτό που είδαμε από την εμπειρία και την πρακτική τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι καταναλωτές δεν κέρδισαν τίποτα και οι αγρότες, ο παραγωγικός τομέας δηλαδή, υπέστησαν τις επιπτώσεις κανόνων που κατέστρεψαν κάθε δυνατότητα συλλογικής διαπραγμάτευτης. Εγώ θυμάμαι ότι παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια μπορούσαμε να κάτσουν οι διάφορες οργανώσεις παραγωγών ε, στο ίδιο τραπέζι με την βιομηχανία για να υπάρξουν κάποιες συμφωνίες για ελάχιστες τιμές χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωστόσο αυτό και Αυτό νομίζω είναι και ο στόχος, να καταστραφεί η διαπραγματευτική μας ικανότητα εξ ολοκλήρου και να παραμείνουμε απροστάτευτοι, τροτοί, ευάλωτοι στα χέρια του, της βιομηχανίας. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε συλλογικές συμφωνίες, αλλά οι βιομηχανίες τα μεταξύ τους. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες καταγγελίες στο Ισπανικό κράτος, για παράδειγμα, που οδήγησε στην επιβολή προστήμων σε γαλακτοβιομηχανίες, για παράδειγμα. Αλλά εν τέλει ε, τα πρόστιμα τα πληρώνει ο παραγωγικός τομέας, γιατί όταν εισπράττονται από επιχειρήσεις, εν τέλει οδηγούν σε μείωση των τιμών των προϊόντων μας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προχωρήσουμε προ μια κατάσταση όπου επανέρχεται το δικαίωμα στην συλλογική διαπραγμάτευση, το δικαίωμα σε συμφωνία για ελάχιστες τιμέ, ακόμα δε και να επιτρέπεται στι κυβερνήσει να λειτουργούν ε, ως διαμεσολαβητές σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία. Αυτό που συμβαίνει σε άλλου ε, εργασιακούς χώρους. Αυτή τη μικρή σκέψη θέλω να κάνω, τις μικρές σκέψεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Δεν ξέρω ε, σε τι βαθμό αποτελεί συζήτηση αυτό που κάνουμε, διότι γίνεται τακτικά αυτό. Ε, κάθε φορά λέμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, αλλά τελικά βλέπουμε ότι η κατάσταση συνέχεια επιδεινώνεται. Να σας πω κάποια νούμερα. Τα 10 μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ ε, αντιπροσωπεύουν το 40% της αγοράς. Σε πολλές χώρες είναι το 75% της αγοράς. Δεν έχουμε ανταγωνισμό. Όπως επιθυμεί η κοινή οργάνωση αγοράς σε διάφορους τομείς. Στο γάλα προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τους παραγωγούς με τις προτάσεις μας που κατά τη γνώμη μας ε, δεν αρκούσαν αλλά αποτελούσαν μια προσπάθεια. Όταν λοιπόν ένας γεωργός δεν έχει τη ε, δυνατότητα να πειράσει την αγορά διότι υπάρχει μόνο ένας αγοραστής, ε, τότε δεν υπάρχει ε, ανταγωνισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν τους παραγωγούς, θα πρέπει να τους δώσουν δικαιώματα, διότι δεν μπορούν στον τομέα του γάλακτος να πούν ότι θα απεργήσουμε. Αυτό δεν επιτρέπεται καν στους γαλακτοπαραγωγού στη Γερμανία, διότι αυτό αντίκειται στην νομοθεσία για τα καρτέλ. Και άλλωστε θα πρέπει να απορρευτεί το γάλα ε, αν γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένω λοιπόν εναγωνίως την πρόταση της Κομισιόν. Και συνάδελφος συνάδελφο πριν τρία χρόνια υπέβαλε πρόταση από την οποία εφαρμόστηκαν πολύ λίγα. Κυρία Επίτροπε, λοιπόν, δεν μου αρκούν οι προτάσεις σας. όμορφα λόγια σε μια θεωρητικά ελεύθερη αγορά που για τους, αγορούς, που για τους παραγωγούς όμως ε, δεν είναι ε, ε, τόσο ελεύθερη. Και όλοι γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση στην αγορά του γάλακτος. Μιλάμε για μια αρρύθμιστη αγορά, μια απελευθερωμένη αγορά με δυνατότητα εξαγωγής σε διεθνές επίπεδο, αλλά οι υποσχέσεις αυτές δεν εκπληρώνονται στην αγορά αυτή και αυτό δεν ισχύει μόνο στον τομέα του ελαιόλαδου, αλλά ισχύει και στο γάλα. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε πάλι με τις βασικές αρχές και νομίζω ότι αυτό που είπε ο Άλμπερτ Τεντές ε, παραβλέπει το πρόβλημα. Διότι το θέμα δεν είναι η φορολογία, είναι τα δικαιώματα των παραγωγών και είναι χρέος μας να ενισχύσουμε τους παραγωγούς. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και η Κομισιόν να κάνει κάτι. Καλό θα ήταν να είμαστε λίγο περισσότερο αισιόδοξοι, αγαπητέ συνάδελφε. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα και χαίρομαι διότι υπάρχει Επιτροπή Ανταγωνισμού και Επιτροπή Γεωργίας στο Κοινοβούλιο γιατί αυτά τα δύο αντίκυνται μεταξύ τους. Όποιος είναι επικεφαλής της αλυσίδας τροφίμων, είτε είναι μια εθνική κυβέρνηση, είτε είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να ικανοποιήσει δύο στόχους που είναι αντιφατικοί μεταξύ τους. Από τη μία πρέπει να διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε ζει υπό τον έλεγχο ε, του φορέα αυτού έχει να φάει σε εφικτές τιμές, προσβάσιμες τιμές και από την άλλη ότι υπάρχει μια κάποια ασφάλεια τροφίμων. Δηλαδή δεν, ότι ο λαός δεν εξαρτάται πλήρως από τις εισαγωγές και ότι μια κάποια εσωτερική παραγωγή είναι βιώσιμη. Ε, αυτά τα δύο είναι πολύ δύσκολο να συμβιώσουν και να συνάδουν. Στο Ενωμένο Βασίλειο έγινε μεγάλη προσπάθεια κάτι να γίνει. Και θέλω να μιλήσω γι' αυτό γιατί είμαι γνώστης στον τομέα των ε, αυγών, τον οποίο γνωρίζω, ε, όπως ξέρετε ε, τα τέσσερα μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ είναι αυτά που διακινούν τη μεγαλύτερη ποσότητα των τροφίμων και ε, απέκτησαν τελικά τέτοια ισχύ που συνεχώς οι αυγοπαραγωγοί έκαναν διαρθρώσεις, συγχωνεύσεις ε, και το καθεξής αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό. Όταν το Deans και το Stonegate συγχωνεύτηκαν, τότε είχαν μια ευκαιρία να γίνουν ισχυροί και θα μπορούσαν να θέσουν στο στόχαστρο οποιαδήποτε αλυσίδα σούπερ μάρκετ και δεν μπορούσαν ε, τα σούπερ μάρκετ να τους πούν δεν μας ενδιαφέρεται πια θα πάρουμε απαλού γιατί ήταν υπερβολικά ισχυροί. Όμως η Βρετανική Επιτροπή Ανταγωνισμού τελικά δεν επέτρεψε τη συγκέντρωση, τη συγχώνευση αυτών των δύο μεγάλων εταιριών αυγοπαραγωγής ε, προς του Βρετανού καταναλωτή υποτίθεται. Δηλαδή ε, τους εξανάγκασαν να αποσυγχωνευθούν. Είχαν, συγχωνευθούν για να, ε, είχαν συγχωνευτεί για να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ε, και τελικά το πρόβλημα ήταν ότι αποσυγχωνεύτηκαν, ακυρώθηκε αυτή η συγχώνευση και οι τιμές εκτοξεύθηκαν τελικά ε, για τους καταναλωτές, αλλά... Ε, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν καλές για τους παραγωγούς. Μια συμβολεακή τιμή μπορεί να είναι καλή παρά μόνο ε, ε, όταν ε, το κοπάδι για παράδειγμα ε, ε, φεύγει νωρίτερα. Π.χ. ένα κοπάδι πρέπει να κρατηθεί 72 εβδομάδες αλλά αν θέλει ο παραγωγός να διατηρήσει την τιμή του συμβουλέου πρέπει να το διώξει στις 68 εβδομάδες. Αυτό το δίλημα του θέτουν ενώπιον του οι αγοραστές. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε. Και να σας μιλήσω και για την Βραζιλία. Είχε έρθει ο Βραζιλιάνος Υπουργό Γεωργίας. Είναι μια χώρα που τα πάντα τα κάνουν σχεδόν καλύτερα από εμάς. Και αν υπάρχει αληθινός ανταγωνισμός ε, τότε με το δικό του ζωικό κεφάλαιο θα πλημμυρίσουν τη δική, τους, τη δική μας αγορά. Ωραία, οι Ευρωπαίοι θα αγοράσουν φτηνά κρέατα. Ναι, αλλά αν οι Βραζιλιάνοι μας κλείσουν τη στρόφιγγα για πολιτικούς λόγους, γιατί μπορεί να τους έχει χτυπήσει μια καταιγίδα σε κάποια δεδομένη ε, χρονική στιγμή, τι θα γίνει με τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Εν πάση πτώση είναι λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα αυτά και χαίρομαι που πρόεδρε συγκαλέσατε αυτή τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ναι. Το θυμόμαστε όλοι. Ε, θυμόμαστε όλοι αυτή τη συνάντηση με τον Βραζιλιάνο Υπουργό Γεωργίας. Την είχαμε πρόσφατα αυτή τη συνάντηση. Ας περάσουμε τώρα στις παρεμβάσεις των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω πολλούς εγγεγραμμένους στο κατάλογο των ομιλητών. Πολλοί θέλουν να πάρουν το λόγο. Να δώσω 1,5 λεπτό στον κάθε ένα. Ο κύριος Νταντέγκη είναι εισηγητής για το θέμα της μεταρρύθμισης Merci, euh, Monsieur le Président. Για το θέμα της μεταρρύθμισης της κοινή γεωργικής πολιτικής, ο κύριος Νταντά. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε. Κυρία και κύριοι ε, Επίτροπε, χαιρόμαστε ιδιαίτερως που είστε εδώ για να μιλήσετε για το περίπλοκο ζήτημα του ανταγωνισμού. Ίσως είναι αναγκαίο να υπενθυμίσουμε τη βούληση του νομοθετή κατά την τελευταία μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Η δημόσια εξουσία δεν ήθελε πλέον να ασχοληθεί με τη ρύθμιση των αγορών. Στις περισσότερες χώρες θεωρήσαμε λοιπόν σκόπιμο να ενισχύσουμε το δικαίωμα των αγροτών και των παραγωγών να οργανώνονται, να οργανωθούν μπορούν για να αντιμετωπίσουν αγοραστές και άλλα, άλλους κλάδους που είναι πολύ πιο ισχυροί. Δεν έχετε απέναντί σας την Google. Έχετε μία μάζα αγροτών που ξέρουν πώς να παράγουν ξέρουν τον νόμο που διέπει την παραγωγή αλλά δεν ξέρουν καθόλου το εμπορικό δίκαιο που ε, διέπει την ίδια τους την παραγωγή. Να ενισχύσουμε λοιπόν την δύναμη όλων αυτών των κλάδων της ε, γεωργίας είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Δίνουμε έτσι σε αυτή τη μάζα αγροτών και παραγωγών ένα αληθινό δικαίωμα εμπορικής έκφρασης, να εκφραστούν και εμπορικά. Αυτό, τους δίνουμε, αυτό το δικαίωμα τους δίνουμε όταν τους επιτρέπουμε να οργανώνονται αυτό που επιθυμήσαμε με τις κατευθυντήριες γραμμές που σας ζητήσαμε είναι το εξής. Να υπάρχουν εγχειρίδια και ζητώ συγγνώμη για αυτή την έκφραση, να δημοσιευθούν εγχειρίδια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε όλοι οι αγρότες, όλοι όσοι δεν έχουν ένα στρατό νομικών επιστημόνων από πίσω τους όπως έχουν οι μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις να μπορούν οι αγρότες να δράσουν μαζί στο σύνολο των χωρών από όποια χώρα και προέρχονται με όσο το δυνατό πιο ομοιόμορφο τρόπο. Η δουλειά του εισηγητή έχει δείξει ότι πράγματι από τη μία χώρα στην άλλη οι πρακτικές είναι τελείως διαφορετικές από πλευράς ε, των εκάστοτε αρχών ε, ρύθμισης θεμάτων ανταγωνισμού οι οποίες όμως αρχές βασίζονται στα ίδια ευρωπαϊκά κείμενα. Θέλουμε λοιπόν να σεβαστούμε τις ευρωπαϊκές αξίες και να επιτρέψουμε στους αγρότες πραγματικά να λειτουργήσουν. Ε, και θα ήθελα να σα θέσω το εξή ερώτημα. Εδώ και 50 χρόνια είναι σαφές ότι το, δίκαιο του ανταγωνισμού δημιουργήθηκε προς το συμφέρον του καταναλωτή για να μειωθούν οι τιμές. Στην Ευρώπη έτσι όπως έχει σήμερα δεν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση κατά την οποία το δίκαιο του ανταγωνισμού ε, λαμβάνει επαρκώς υπόλοιπη υπόψη τα θέματα της υπεράσπισης της απασχόλησης. Γιατί όταν θέλουμε πάντοτε να βρίσκουμε φτηνά προϊόντα σε φτηνές τιμές, πάντοτε υπάρχει κάποιος που πουλάει φτηνότερα και φτηνότερα και φτηνότερα από ότι εμείς που το παράγουμε. Πάντοτε θα υπάρχει κάποιος παραγωγός στον πλανήτη σε αυτή τη φρενήρη κούρσα. Όσο λοιπόν αγοράζουμε το όλο και πιο φτηνά, τόσο περισσότερες θέσεις απασχόλησης χάνουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το δίπολο όχι μόνο πολίτη πολίτη καταναλωτή αλλά και πολίτη μισθωτού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκαρσία. Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας ότι ο κλάδος πρέπει να κερδίσει χρησιμοποιώντας περισσότερη, περισσότερο ανταγωνισμό και καινοτομία. Αυτό είναι και ο στόχος της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ. Ωστόσο, εδώ λείπουν κάποια πράγματα. Πώς εφαρμόζεται η διαπραγμάτευση των συμβάσεων αναφέρεται. Δεν εξετάζεται ωστόσο η εναρμόνιση του ανταγωνισμού αυτή καθ' αυτή. Εγώ προερχόμαι από την Ισπανία όπου η αρχή ανταγωνισμού είναι αρκετά πρωτότυπη σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη όπως τη Γαλλία. Ο τομέα των αγροδιοτροφικών προϊόντων υπέστη πολλά στη χώρα μου. Γι' αυτό πρέπει να υπάρξει μια ομοιογενή ερμηνεία των κανόνων ανταγωνισμού στον ε, τομέα των προϊόντων διατροφής σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, δεν μπορούμε, άλλο θέμα αυτό, να θεωρήσουμε υπεύθυνου τους ε, γεωργούς για την αποτελεσματικότητα των, ε, του κλάδου. Δεν μπορεί να είναι αυτοί μόνο υπεύθυνοι για τις προσιτές τιμές στους καταναλωτές. Η διανομή, η μεταποίηση δεν παίζουν αυτές ένα σημαντικό ρόλο όλοι οι κρίκοι της ε, αλυσίδας διατροφής παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Για τους τρεις κλάδους που αναφέρεται, αυτό που με ανησυχεί είναι περισσότερο είναι το ελαιόλαδο. Γιατί το να ζητήσουμε, όπως αναφέρεται, ότι ένα, το μεγαλύτερο ποσοστό ελαιολάδου των οργανώσεων παραγωγών να είναι ε, εμφιαλωμένο ή μετακίνηση ή μεταφορά να γίνεται από κοινού από τις οργανώσεις παραγωγών δεν είναι ρεαλιστικό. Αν ξέρετε τον κλάδο του ελαιολάδου στην Ισπανία, οι κανόνες αυτοί που σα πω δεν εφαρμόζονται. Τουλάχιστον δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε εμά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μποβέ. Πρόεδρε. Επίτροποι. Ο συνάδελφος θύμισε ότι το 2012 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπεψήφισε μία έκθεση για την καλύτερη κατανομή της υπεραξίας της αλυσίδας διατροφής μεταξύ των αγροτών, της ε, μεταποίησης και της διανομής. Έκθεση που ψηφίστηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία στηριζόταν σε συγκεκριμένα δεδομένα ότι τα τελευταία 15 χρόνια η μερίδα της γεωργικής πραξίας που έπαιρναν οι γεωργοί πέρασε από το 30% σε κάτω του 20% σήμερα. Δηλαδή οι γεωργοί σε 15 χρόνια έχασαν ένα μεγάλο κομμάτι των χρημάτων τους προς όφελος των μεταποιητών και της μεγάλης διαμονομής ιδίω. Το θέμα λοιπόν του ανταγωνισμού που αναδείχθηκε από τον Μισελ Νταντάν προηγουμένως ε, λέει πολύ σαφώς τα πράγματα. Πρέπει να ξαναμοιράσουμε την γεωργική υπεραξία σε όλο τον κλάδο. Δύο παραδείγματα θα σας δώσω. Πρώτον, όταν μειώθηκε η τιμή του γάλακτος το 2009, δεν είδαμε μείωση της τιμής του γάλακτος στη διανομή. Αυτό δείχνει ότι τελικά δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Κανονικά θα έπρεπε να κερδίσει και ο καταναλωτής. Δεν έγινε. Δεύτερο παράδειγμα που πραγματικά σοκάρει ο παραγωγός οπροκυπευτικών. Όταν οι παραγωγοί των οπροκυπευτικών οργανώθηκαν, ΜΑΤΕ στη Γαλλία, ε, καταγγέλθηκαν από την Ευρώπη διότι έκαναν οργάνωση για συλλογική πώληση και είπαν ότι αυτό είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Νομίζω ότι εδώ πραγματικά ε, πάμε λάθος, σε λάθος δρόμο. Αυτή τη στιγμή η παραγωγή δεν είναι η απειλή, είναι, είναι διασπασμένη. Η απειλή είναι οι, μεγάλες, ε, οι μεγάλοι όμιλοι ε, Μεταποίηση και διανομής. Όσο μεγαλύτερη συγκέντρωση γίνεται στον χώρο της διανομής και οι αλυσίδες, ε, και οι αλυσίδες τροφίμων ε, συγκεντρώνονται, δεν παραπέμπονται για στρέβλωση του ανταγωνισμού, αλλά τους δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε όχι μόνο στους τρεις κλάδους που αναφέρεται αλλά σε όλη τη γεωργία διότι και η μεταρρύθμιση και η, έκθεση για τον, την ενιαία κοινή οργάνωση αγοράς δεν γίνονται λόγος για όλα τα θέματα. Τα για παράδειγμα πρέπει να μπουν εξ αρχής στη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ την κυρία Βεστάγκερ για την παρουσία της εδώ. Είναι καλό πράγμα για τη δουλειά μας. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Χόγκαν. Συχνά τον βλέπουμε βέβαια. Συμφωνώ με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν. Απλώς ήθελα να ρωτήσω γιατί αναφέρονται αυτά τα προϊόντα και όχι άλλα. Το γάλα, για παράδειγμα, το είπαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Επίσης, να ρωτήσω, υπάρχουν νέες καθοδηγητήριες γραμμές. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Η πλαισίωση των ε, συνεταιρισμών θα αναφέρεται θα υπάρχει μνήμα ότι οι συνεταιρισμοί θα θεωρούνται ως οργανώσεις παραγωγών και άλλα θα έχουν τους ίδιους ανταγωνι... το... τις ίδιες εξαιρέσεις σε θέματα ανταγωνισμού, διότι το κείμενο δεν είναι σαφές στα σημεία αυτά. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους Επιτρόπους και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρεσε. Ρωτώ την Επίτροπο Φεστάγκερ το εξή. Με χαρά σας άκουσα να λέτε ότι ο γεωργικός τομέας προφανώς αντιμετωπίζει προκλήσεις και από πλευρά συνεισφοράς και από πλευρά αγοραστών. Χαίρομαι που το λέτε, διότι θεωρώ ότι καταλαβαίνετε ότι οι αγρότες είναι αυτοί που παίρνουν την τιμή που τους παρουσιάζουν και δεν διαμορφώνουν την τιμή που θέλουν. Υπάρχουν και άλλες απειλές, όπως είναι οι πρακτικές για το αθέμητο εμπόριο. Ο κύριος Νταντά έχει κάνει τεράστια δουλειά ε, για τα θέματα του ανταγωνισμού εγώ ασχολούμαι με την εφοδιαστική αλυσίδα. Επανειλημμένως η δική μας Επιτροπή έχει ψηφίσει υπέρ της ισχυρότερης θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει πιο ισχυρή θέση. Είναι εξωφρενικό το κάθε κράτος μέλος να λειτουργεί διαφορετικά, να κάνει το δικό του, προσπαθώντας η εφοδιαστική αλυσίδα να λειτουργήσει καλύτερα από τον παραγωγό μέχρι τα δικαιώματα του καταναλωτή. Δεν υπάρχει καμία διαφάνεια για τη διαμόρφωση των τιμών. Είναι μια μαύρη ε, όλο αυτό. Όλοι είμαστε καταναλωτές, όλοι αγοράζουμε τρόφιμα, αλλά δεν κατανοούμε τις, τους μηχανισμούς διαμόρφωσης της τιμής, τις ειδικέ προσφορές και από πλευράς αηφορίας δεν γνωρίζουμε τις συνέπειες της ατελούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Έχω παρακολουθήσει όλους τους επιτρόπους από την εποχή του επιτρόπου Φίσλερ και πιο πριν. Ο, καθένας, ο κάθε επίτροπος Γεωργίας έχει τη δική του μεταρρύθμιση. Κάθε φορά έχουμε λιγότερο προϋπολογισμό, έχουμε περισσότερες απαιτήσει από τους αγρότες και τους λέμε πηγαίνετε στην αγορά να δοκιμαστείτε. Όμως η αγορά είναι ατελής, δεν είναι τελεία και θα πρέπει η Επιτροπή να αναλάβει δράση. Γνωρίζετε την επιστολή που σας εστάλει για να σας καλωσορίσουμε στη θέση της Επιτρόπου του Ανταγωνισμού. Μία από τις λέξεις στη γνωστή επιστολή είναι ότι ελπίζουμε ότι θα κάνετε ένα φρέσκο ξεκίνημα. Είναι η τρίτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έχω παρακολουθήσει αυτή την πρωτοβουλία για την εφοδιαστική αλυσίδα, ε, την αγροδιατροφική αλυσίδα. Έχω παραστεί σε όλες τις συνεδριάσεις, με όλους τους εταίρους, με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Πάρα πολύ ωραία λόγια έχω ακούσει χρόνια τώρα, αλλά εν πάση δεν έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οριστική δράση για το θέμα αυτό και πρέπει να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβουμε υπόψη το θέμα της αηφορίας. Αυτή η ιδέα των φτηνών τροφίμων χωρίς ε, καμία ε, σκέψη για την αηφορία ε, της παραγωγής δεν μας φτάνει, δεν είναι αρκετά καλή, δεν φτάνει αυτό το πράγμα και οι άλλοι συνάδελφοι σας παρουσιάσαν συγκεκριμένα παραδείγματα για την παράξενη στάση των αγροτών σε σχέση με τον λιανοπολιτών. Έχουμε επιτρέψει αυτή την κατάσταση να συμβεί και να διαιωνιστεί. Ως καταναλωτές ε, επιλέγουμε ανάμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε πραγματικά μια αληθινή, ε, πραγματική επιλογή ε, μπροστά μας και πρόεδρε θα σας παρακούσω και δεν θα μιλήσω μόνο ένα μισή λεπτό. Είναι μια μοναδική ευκαιρία. Έχουμε μπροστά μας δύο επιτρόπους, δύο πολύ σημαντικά χαρτοφυλάκια που έχουν αντίκτυπο ε, στη δουλειά μας. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει σοβαρά την έκθεσή μας, να ακούσει, να διαβάσει τα περασμένα ψηφίσματα, να διαβάσει τις εκθέσεις της Επιτροπής μας και βάσει να κάνει το παν για διαφάνεια και για καλύτερη αντιμετώπιση και των καταναλωτών και των αγροτών. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ε, ο ρόλος μου είναι κάπως δύσκολος, αλλά πρέπει να τον παίξω. Και γι' αυτό οφείλω να σας διακόψω. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να μην μιλήσω τόσο πολύ όσο η κυρία Μαγκίνες. Καταρχάς να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους για την παρουσία τους εδώ. Είναι πολύ σημαντικό που είστε και οι δύο εδώ παρόντες ο Επιτρόπος ε, Γεωργία συχνά έρχεται να μας δει και τον ευχαριστώ και έχουμε και την Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό, η οποία έρχεται λιγότερο συχνά και την ευχαριστώ ιδιαίτερω για την παρουσία της εδώ. Γνωρίζω καλά την κατάσταση και τα προβλήματα στην αγορά, αγορά του ελαιολάδου. Είμαι από την Ανδαλουσία, μια περιφερεια όπου το ελαιόλαδο έχει καθοριστική σημασία ε, σε βάθο χρόνου, όχι πρόσφατα, και στις περισσότερες ε, κοινότητες ε, και Δήμου. Έχουμε κοινή οργάνωση αγορα σε πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά Συμφωνώ απολύτως με τους προλαλήσαντες. Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση. Το πρόβλημα με το ελαιόλαδο είναι ότι κάθε χρόνο ο όγκος της παραγωγής διαφέρει ιδιαιτέρως. Έχουμε χρονιές όπου έχουμε πολύ μεγάλη παραγωγή, πέφτουν οι τιμές ε, λογικά και έχουμε άλλα χρόνια όπου έχουμε πολύ μικρότερη παραγωγή γιατί το κλίμα επηρεάζει την παραγωγή και ο ελαιώνας είναι κάτι το μετάβολο και το τυχαίο και γι' αυτό έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές στην ε, παραγωγή. Και πολύ συχνά αυτό δεν γίνεται κατανοητό. Σε ορισμένες χρονιές ζητούν ε, οι ελαιοκαλλιεργητές ε, την ιδιωτική αποθήκευση και την άλλες χρονιές ζητούν συγκεκριμένες τιμές. Θα σας διαβιβάσω γραπτός ορισμένες γνωμοδοτήσεις για το ελαιόλαδο πιο συγκεκριμένα. Ε, προς το παρόν όμως θέλω σήμερα εδώ να σας πω ότι για τη δέσμη μέτρων για το γάλα και τα γαλακτοκομικά ε, θα ψηφίσουμε τη σχετική έκθεση εντός ολίγου. Να σας πω ότι είχαμε υποχρεωτικές αιτήσει συμβάσεις, συμβόλαια στη χώρα μου ε, κατά κύριο λόγο και δεν λειτουργούν. Οι αγρότες συνεχίζουν να παίρνουν τα ε, πάρα πολλές ε, χαμηλές τιμές, πάρα πολύ χαμηλές τιμές για τα προϊόντα τους. Στον τομέα των οποροκυπευτικών έγινε οργάνωση παραγωγών οποροκυπευτικών που αποθήκευσαν μεγάλες ποσότητες, ούτε αυτό λειτουργήσε. Άρα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ερμηνείας των κανόνων του ανταγωνισμού και ε, στην χώρα μου, στην Ισπανία, ε, είναι κάτι που εφαρμόζεται συνεχώς σε άλλες χώρες όχι. Ολοκληρώνω Πρόεδρε λέγοντας στην Επίτροπο, στον Επίτροπο κύριο Χόγκαν ότι εμείς αγωνιζόμαστε για έναν αγροτικό κλάδο πιο δίκαιο, πιο αηφόρο και πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί με να είναι πιο αηφόρος και πιο ανταγωνιστικός, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα περισσότερο δίκαιος. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Κυρίε και κύριοι, δεν θα έχουμε αρκετό χρόνο και από τη στιγμή που θέλουμε να ακούσουμε τις απαντήσεις των Επιτρόπων, παρακαλώ να είστε σύντομοι. Επόμενος ομιλητής. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι καλό το ότι βρίσκονται εδώ οι δύο επίτροποι. Είναι πολύ σημαντική και η καλή συνεργασία. Δεν ε, αρκεί μόνο η παραγωγή, πρέπει να ισχύουν και οι καλές συνθήκες ανταγωνισμού για τους γεωργούς. Συζητάμε τώρα τις κατευθυντήρες γραμμές. Συζητάμε τι μορφή έχει μια ισορροπημένη σχέση ανάμεσα στους παραγωγούς. Υπάρχουν πολλές πτυχές όπου δεν υπάρχουν δίκαιες συνθήκες που συνδέονται με τα διάφορα μέτρα. Μπορεί στο πλαίσιο του ίδιου μέτρου ένας να λαμβάνει 70 ευρώ, άλλος 100%. Είναι πολύ δύσκολο να ε, δει κανεί σε τι είναι δίκαιο. Ο κύριος Χόγκαν ε, ασχολείται με το θέμα. Από την άλλη, θα ήθελα να θίξω και ένα άλλο πρόβλημα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι το οποίο δεν έχει λογική εξήγηση. Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί ε, δεν επιτρέπεται να καλλιεργηθούν, μπορούν όμως ε, να εισάγονται. Κύριε Επίτροπε, βρίσκεται ότι είναι καλό να έχουμε αυτά τα διπλά μέτρα. Δηλαδή, ή δεν είναι ενια οι οργανισμοί αυτοί και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να τους καλλιεργούμε και να τους εισάγουμε, ε, ή θα πρέπει να επιτρέπονται. Και επίσης, όσον αφορά την αγορά γάλακτος, ε, επικρατούν πολύ δύσκολες συνθήκες αυτή τη στιγμή και έχετε να παίξετε σημαντικό ρόλο όταν βλέπουμε τι ισχύει εκεί. Και έχουμε και την κατάσταση απέναντι στη Ρωσία. Κύριε Πρόεδρε, ολοκληρώνω. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ε, είναι η Ρουμανία έχουν πλημμυρίσει από φτηνά ε, γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία πολλούνται με τιμές dumping, πολλούνται με, ε, για ένα ευρώ τη στιγμή που έχουν στοιχήσει δύο ευρώ. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Γιάρε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικός ο ανταγωνισμός. Δύο σύντομες παρατηρήσεις. Ε, καταρχάς βρίσκω καλό το ότι δεν συζητάμε σήμερα σχετικά με τη διαμόρφωση των ε, τιμών διότι έτσι δεν θα φτάσουμε στο πραγματικό πρόβλημα. Ωστόσο σημαντικό είναι αυτό που υπόθηκε. Θα πρέπει να έχουμε ολοκλήρωση της κοινή αγοράς ε, και να φροντίσουμε να μην εμποδίσουμε την ολοκλήρωση αυτή με τις αποφάσεις μας. Υπάρχουν διαφορές ε, στις άμεσες πληρωμές οι οποίες όμως ε, δεν ε, δικαιολογούνται. Ο κύριος ε, Ντόρφαν ίσως να μπορεί να το εξηγήσει αυτό περαιτέρω. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε με πιο δικαίο τρόπο τις άμεσες πληρωμένες. Επίσης, όσον αφορά την διαμόρφωση των τιμών, έχουμε λίγους παραγοντές στις αγορές, έχουμε τα ε, τα σούπερ μάρκετ δεν χρειάζεται καν να, να συνοηθούν μεταξύ τους, είναι τόσο λίγοι, αλλά έτσι πέφτουν οι τιμές. Πώς μπορούμε λοιπόν να έχουμε σωστή διαμόρφωση των τιμών, ώστε να επιτρέπεται οι γεωργοί να συνεννοούνται μεταξύ τους, διότι πρέπει να έχουν διασφάλιση κάποιων ε, ελάχιστων ε, τιμών. Και έχουμε σε κάποια προϊόντα, κάποια μέτρα τα οποία δεν έχουμε σε άλλα. Θα πρέπει να ασχοληθούμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Oui, merci, Alors, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το να διευκολύνουμε τους κανόνες να οργανώνονται για να αντιμετωπίσουν την διανομή και τη μεταποίηση είναι καλό. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή όλοι οι κλάδοι έχουν ε, προβλήματα στρέβλωσης από τις μεγάλες αλυσίδες διανομής κατηγορώντας ότι πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω. Άκουσα ένα συνάδελφο να αναφέρει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στους γεωργούς, να γίνει μια πιο δίκαιη γεωργία. Πώς αυτά θα γίνουν κύριε Χόγκαν, ε, ο ανταγωνισμός σε ένα πλαίσιο ακραίου φιλευθερισμού οδηγεί σε συγκέντρωση των εκμεταλλεύσεων και άρα στην εξαφάνιση των μικρών εκμεταλλεύσεων. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε και στο γαλακτικό τομέα και στην κοινοτροφία. Οι γεωργοί ε, κάνουν συγκέντρωση για να επιβιώσουν. Δεν είναι επιλογή, είναι συνέπεια του συστήματος. Αυτή η προοπτική έχει επιπτώσεις και στην ύπεθρο σε ό,τι αφορά την απασχόληση των ε, κατοίκων της, της επαρχίας και την απερίμωση της επαρχίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος. Πρόεδρε. Συζητήσαμε το θέμα αυτό πλιστάκης θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο. Πέραν των συζητήσεων πρέπει να κάνουμε και κάτι. Το ότι είναι σήμερα στη συνάντησή μας δύο επίτροποι είναι μαρτυρία το ότι έχουμε επίγνωση το πρόβλημα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Οι γεωργοί σε πολλούς κλάδους δεν μιλούν για προοπτικές, προσπαθούν να επιβιώσουν. Στις βαλτικές χώρες για παράδειγμα η τιμή, οι τιμές που εισπράττουν οι γεωργοί σήμερα είναι μισές από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Σκέφτονται όλοι να φύγουν από τον κλάδο τους και να πάνε σε έναν άλλο κλάδο. Αν ο κόσμος δεν μείνει στο ο κόσμος δεν μένει στο χώρο της γεωργίας, το βλέπουμε αυτό. Ε, στην ουσία χρησιμοποιεί τη γεωργία για πρώτες Ο έμπορος επιλέγει ό,τι νομίζει καλύτερο. Ο γεωργός αντιμετωπίζει συνεχώς τον κίνδυνο της ε, πτώχευσης. Γιατί του λέει ο έμπορος ότι άμα δεν μειώσει τις τιμές θα πάρουμε από αλλού. η εναλλακτική λύση είναι να δώσουμε ξανά εξουσίες στα κράτη-μέλη για να προστατεύσουν αυτά τις αγορές του. Ο κύριος Ντελάιερ, η κυρία Ντελάιερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ε, επιτρόπους την προσία τους. Να σας πω τη δική μου εμπειρία ως ε, ε, παραγωγού και εμπόρου προκυπευτικών. Εδώ και 25 χρόνια την ίδια δυσκολία αντιμετωπίζω με την αλυσίδα διανομής. Μου επιβάλλουν συσκευασίε που δεν μπορώ να επιλάξω. Δεν μπορώ να διαπραγματευτώ την τιμή του. Δεν μπορώ να εξασφαλίσω αν έχουν ποιότητα υγειονομικού χαρακτήρα. Ε, Δημιουργώντα προβλήματα στην εκμετάλλευσή μου από μεταφορά ιών που προέρχονται από τρίτες χώρες ε, προς την Ευρώπη. Θα ήθελα ως ε, παραγωγός να προστατεύουμε καλύτερα από την Κομισιόν έναντι αυτών των καταχρηστικών πρακτικών. Πρέπει σήμερα να δουλέψουμε ουσιαστικά για τον το ανταγωνισμό, για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης που ε, βλάπτει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά και την διαχείριση κρίσεων καθώς και την προσαρμογή της προσφοράς και της ζήτησης και τον καθορισμό των τιμών. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ως γεωργοί να υφιστάμεθα κανόνες ανταγωνισμού που δεν είναι καθόλου προσαρμοσμένοι σε παραγωγές που είναι τυχαίες ε, λόγω κλιματικών φαινομένων. Βλέπουμε τις επιπτώσεις του κλίματος στην παραγωγή και στην κατανάλωση κάθε ζημία δεν, καμία ζημία δεν αποζημιώνεται στον γεωργό και σας ε, το λέω αυτό και ως, κατα... και ως γεωργός και ως καταναλώτρια. Ευχαριστώ. Ο κ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα είναι η συζήτηση και χαίρομαι που είναι εδώ οι δύο επίτροποι. Ελπίζω να έχουμε και άλλες τέτοιες συναντήσεις. Συχνά συναντάμε άτομα που δεν βλέπουν καμία σχέση μεταξύ των τροφίμων και της γεωργίας. Ε, πιστεύουν ότι το γάλα έχετε σε μπουκάλια. Δεν σκέφτονται τη γεωργία. Και να το σκέφτονται ωστόσο κάποιοι, εντάξει, δεν είναι σοβαρό πρόβλημα. Όταν το σκέφτεται όμως ένας πολιτικός, αυτό είναι πρόβλημα. Πρόσφατα είχα ασχοληθεί με τη μεταρρύθμιση του κλάδου της ζάχαρης και με το greening αλλά και τα γαλακτοκομικά. Επιβάλλονται στον κλάδο το γαλακτοκομικό εξαιρετικά αυστηρές εξαιρετικά αυστηρά πρόστιμα προς τους γεωργούς αν ξεπεράσουν τις ποσοστώσεις. Αυτό είναι απαράδεκτο. Η πολιτική μας πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να αγοράζουμε τρόφιμα από το εξωτερικό. Θέλουμε να μιλήσουμε για ανταγωνιστικότητα. Η γεωργία, η ευρωπαϊκή γεωργία δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστική δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες, τη Βραζιλία και άλλες χώρες και για λόγους κλιματικούς και για λόγους γεωγραφικούς και στην εσωτερική μας αγορά δεν μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών συχνά οι διαφορές αυτές γίνονται εντονότερες πρέπει να αλλάξουμε πορεία να σκεφτούμε την προστασία της γεωργίας διότι πρέπει η γεωργία αυτή να μπορεί να επιβιώσει. Μετά μόνο θα μιλήσουμε για ανταγωνιστικότητα και ανταγωνισμό. Ευχαριστώ. Um, I start, I'm just wondering... Πριν ξεκινήσω, αναρωτιέμαι όλοι οι Ιρλανδοί μιλάμε ναι, για τέσσερα λεπτά ή αυτό ισχύει μόνο για την κυρία Μακίνες. Μπορείτε να μου απαντήσετε παρακαλώ. Ένα λεπτό είπατε, Άννα Ευρωβουλευτή. Πόσο χρόνο ομιλίας έχουμε, παρακαλώ. Ε, Ενάμιση λεπτό. Η κυρία Μαγκίνες μίλησε περισσότερο γιατί καταρτίζει έκθεση για το θέμα αυτό για την εφοδιαστική αλυσίδα. Ενάμιση λεπτό έχετε παρακαλώ. That's, that's good enough. Εντάξει, Απλά θα ήθελα να πω ότι είμαστε ίσοι, θα ήθελα ε, να έχω την ίδια μεταχείριση παρότι είχα πολλές, πολλές περισσότερους ψήφους από την κυρία Μακίνες. Στο ίντερνετ είδα ε, μια ε, επιγραφή που έλεγε ότι αν φάγατε σήμερα ευχαριστήστε έναν γεωργό. Όχι ευχαριστήστε την Εστλέη ή την Τέσκο και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό διότι χωρίς τους γεωργούς η Τέσκο ή η Νεστέ δεν πρόκειται να ταΐσει τα παιδιά μας. Θα πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε τους ε, γεωργούς και να φροντίσουμε για τη διαβίωσή τους. Και αυτό που κάνουμε είναι ακριβώς το αντίθετο. Σε λίγο δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης και τι θα κάνουμε τότε. Κάτι που θα πρέπει να κάνουμε και νομίζω θα μας βοηθήσει είναι το εξής. Πολλά ακούμε για το δίκαιο εμπόριο, fair trade, αγοράζω τσάι ε, που προέρχεται από τέτοιο εμπόριο και γνωρίζω πολλές ε, νοικοκυρές ε, και νοικοκυριτέ που κάνουν ακριβώς το ίδιο, επιλέγουν τέτοια προϊόντα. Και το κάνουν αυτό επειδή νομίζουν ότι έτσι είναι πιο δίκαιοι. Αλλά νομίζω ότι οι νοικοκυρές και οι νοικοκυρές της Ευρώπης θα πρέπει να γνωρίζουν, για παράδειγμα, όταν αγοράζουν βόλιο κρέα πόσο λαμβάνει ο, ο παραγωγός. Θα πρέπει να ενημερώσουμε το κοινό τους μη γεωργού, ανθρώπους που προέρχονται από οικογένειε σαν τη δικιά μου, που δεν καταλαβαίναμε ε, τι, ε, ποιο ήταν το όφελος των χρημάτων που λαμβάναμε. Το θέμα εδώ πέρα δεν είναι μόνο η γεωργή. Διότι εάν, φύγουν, εάν καταλήψουν οι γεωργοί τις διάφορες περιοχές, δεν θα υπάρχουν πια χρήματα στι περιοχές αυτές. Καταρχά όμω θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει πόσα παίρνει ο γεωργός. Θα ήθελα πολύ να το δω αυτό. Ε, ήδη υποτίθεται ότι έχουμε ανιχνευσιμότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Σκατλή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους ε, δύο επιτρόπους. Ε, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό το ότι βρίσκονται και οι δύο εδώ και ελπίζω η κυρία Βέσταγκερ να έμαθε κάποια πράγματα από τις παρεμβάσεις που ήδη έγιναν. Έχω υποβάλει κάποιες ε, γραπτές ερωτήσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τα λοιπάσματα. Ο κόσμο δεν καταλαβαίνει πώς μειώνονται τα ε, ενεργά συστατικά των διπασμάτων, αλλά αυξάνεται το κόστος. Επίσης, είχα χαλιλογραφία με διάφορες γενικές διευθύνσεις όσον αφορά τον αντίκτυπο και τον έλεγχο στον τομέα του βοηού κρέατος. γενικά ε, θεωρείται ότι υπάρχει καρτέλ και δυστυχώς η Κομισιόν ενώ λέει τα σωστά πράγματα όσον αφορά την δίκαιη αμοιβή των παραγωγών δεν φαίνεται να λαμβάνει την ε, γρήγορη δράση που απαιτείται όταν βλέπουμε διαμόρφωση των τιμών από τους ε, μεγάλους παράγοντες. ενώ το αντίθετο ισχύει όταν οι ε, γεωργικοί συνεταιρισμοί προσπαθούν να πετύχουν δίκαιες τιμές για τα μέλη τους. Το προσωπικό των δύο υπηρεσιών σας ε, λοιπόν θα συνεργαστεί για να διασφαλίσει δίκαιη αμοιβή για τους γεωργούς και ο, ο κόσμος να γνωρίζει ότι όταν ε, αγοράζει γεωργικά προϊόντα μπορεί να είναι βέβαιος ότι και ο γεωργός λαμβάνει δίκαιη αμοιβή. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις, οι παρεμβάσεις των βουλευτών. Έχω την εξής πρόταση. να απαντήσει η Επίτροπος θα δώσουμε το λόγο στους προσκεκλημένους μας. Η Επίτροπος πρώτα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολύ και ευχαριστώ όλους τους ευρωβουλευτές για τις παρεμβάσεις τους. Καταρχάς, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο λόγος που βρισκόμαστε εδώ είναι ότι η Επιτροπή σας ως συνομοθέτης ανέλαβε δράση μαζί με το Συμβούλιο για να επιφέρει αλλαγές. Και αυτό είναι ο λόγος που εκπονήσαμε αυτής τις κατευθυντήρες γραμμές οφείλονται στην αποφασιστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να έχουμε κατά νου. Μπορούν λοιπόν να αλλάξουν τα πράγματα. Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ω προς το θέμα ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι κατευθυντήρε γραμμέ. Συμφωνώ με ε, τον ομιλητή που είπε ότι δεν έχουν ε, όλοι ένα στρατό από δικηγόρου ε, να του βοηθάει να εφαρμόσουν μια σειρά δύσκολων κανόνων. Και αυτός ε, ήταν ένας λόγος που ασχοληθήκαμε με τη διατύπωση, με τα παραδείγματα για να ε, είναι άμεσα εφαρμόσιμοι και χρήσιμοι οι κανόνες. Διότι αλλιώς μπορεί απλά να αποτελούν ωραίες ε, ευκαιρίες στο ράφι, όχι όμως στην καθημερινή ζωή. Αυτός είναι ο βασικός στόχος, να επιτρέψουμε στους γεωργούς σε τρεις συγκεκριμένους τομείς, ε, το βόλιο κρέας, ε, τις αρωτέ καλλιέργειες ε, και το ελαιόλαδο. Να επιτρέψουμε λοιπόν στους αγρότες να οργανωθούν και να έχουν διαπραγματευτική δύναμη την οποία χάνει κανείς αν είναι μόνος του. Ελπίζω να διαβάσετε τις κατευθυντήρες γραμμές έχοντας ακριβώς αυτό κατά νου όσον αφορά απαντήσεις σε κάποια από τα θέματα που τέθηκαν. Καλύπτονται οι συνεταιρισμοί. Οι οργανώσεις παραγωγών μπορούν να έχουν διάφορες νομικές μορφές, εφόσον είναι νόμιμες. Και στην περίπτωση αυτή καλύπτονται. Οι κατευθυντήρες γραμμές θα το καλύψουν αυτό. Βέβαια δεν μπορούμε εμείς να οργανώσουμε τους παραγωγούς, αλλά νομίζω ότι πολλοί Παραγωγή θα ήθελαν να δράξουν την ευκαιρία ώστε να έχουν πιο ισχυρή θέση απέναντι στους ε, αγοραστές. Μετά την οριστικοποίηση αυτών των καθηγητήρων γραμμών θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το σύνολο της ε, αλυσίδας αξίας. Έχουν ε, αναφερθεί η ενέργεια, τα λοιπάσματα και διάφορα ε, και διάφοροι τομείς ε, τους οποίους παρακολουθούμε από κοντά. Η αύξηση των τιμών δεν οφείλονται πάντα σε κατάχρηση δεσπόσες θέσεις. Ε, μπορούν να υπάρχουν σωστοί λόγοι για κάτι τέτοιο, αλλά θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Όπως υπόθηκε, προφανώς Ε, μία μικρή μονάδα ε, πρέπει να δέχεται τις ε, τιμές που υπάρχουν στην αγορά. Θέλουμε λοιπόν να δώσουμε περισσότερη, πιο ισχυρή θέση στον παραγωγό κατά την πώληση. Και επίσης στο πακέτο αυτό βρισκόμαστε σε ένα από τα τελευταία στάδια εξέτασης της κατάστασης όσον αφορά τις συσκευασίες, διότι φαίνεται ότι Υπάρχει δεσπόσα θέση σε κάποιους ε, τομείς ε, που εξηγεί και όλες τις εξελίξεις ε, στην αγορά συσκευασία τροφίμων και μπορεί αυτό να φαίνεται μικρή λεπτομέρεια αλλά για τα προϊόντα είναι πολύ σημαντικό διότι η ποιότητα της συσκευασίας και ο τρόπος παρουσίασης και η επιλογή του παραγωγού σχετικά με το πώς θα παρουσιάσει το προϊόν του είναι πάρα πολύ σημαντικά. Γι' αυτό έχει νόημα να εξετάσουμε και αυτές τις ε, περιπτώσεις που μπορεί, σε, ε, που μπορεί σφαιρικά να μην φαίνονται ότι είναι τόσο σημαντικά, αλλά μπορεί να είναι σημαντικά για τον κάθε παραγωγό. Δεύτερον, ε, έχουμε κάποιες εξελίξεις όσον αφορά την έκθεση για τις αγορές λιανικής και την επισήμανση. Διότι το θέμα είναι αν η επισήμανση αποτελεί εμπόδιο στην καινοτομία. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εξετάζουμε την εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας. Και όσον αφορά την, τον ανταγωνισμό, δεν μας ανησυχούν μόνο οι χαμηλές τιμές. Υπάρχει το θέμα της καινοτομίας και η αποτελεσματικότητα για τον καταναλωτή που αποτελούν λόγοι που ασχολούμαστε με αυτές τις οργανώσεις πολιτών, παραγωγών. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε και άλλα αποτελέσματα πέρα από την διαπραγματευτική θέση όσον αφορά την αποθήκευση, όσον αφορά τη διάθεση στην αγορά. Έτσι μπορούμε να επιτρέψουμε σε μικρούς παραγωγούς να έχουν πολύ πιο ισχυρή θέση. Θα συνεργαστούμε με τη συνάδελφό μας την κυρία Βιενκόφσκα που είναι αρμόδια για την εσωτερική αγορά όσον αφορά τις ε, θεμητές εμπορικές πρακτικές για να δούμε εάν υπάρχει ανάγκη για μια πρωτοβουλία στον τομέα αυτών. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι αυτό που κάνουμε να λειτουργεί και στην πράξη, διότι Σημαντικό είναι στους τρεις αυτούς τομείς, στο βόλιο κρέας, τις αρωτρές καλλιέργειες και το ελαιόλαδο, να δούμε εάν θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες, νέες δυνατότητες. Και ακριβώς γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να λαμβάνουμε και από εσές πληροφορίες σχετικά με το εάν λειτουργούν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμέ όπως είχατε προβλέψει εσείς ως νομοθέτης πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, διότι στόχος μας είναι να έχουμε κάτι άμεσο, συγκεκριμένο και χρήσιμο ακόμα και για ανθρώπους που δεν έχουν ε, μια στρατιά δικηγόρων στη διάθεσή τους. Η τελευταία μου παρατήρηση είναι ότι ελπίζω να λειτουργήσουν οι κατευθύνσεις γραμμές και ε, για τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού, ώστε να έχουμε ε, ορθή εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών και να συμβάλλουμε ακόμα περισσότερο στη διαμόρφωση συνθήκων ίσου ανταγωνισμού. Διότι ακούσαμε πολλές παρατηρήσεις σήμερα σχετικά με το ε, πόσο διαφέρει η θέση των γεωργών ανάλογα με την ε, χώρα και τον τομέα που δραστηριοποιούνται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση και επίτροπε ο κ. Χόγκαν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Σωστά είπε η συνάδελφος κ. ότι κατάλαβε πάρα πολλά από αυτά που παρουσιάστηκαν σήμερα και την ευχαριστώ γιατί εγώ ξέρω να συζητώ με τους ανθρώπους εδώ, δεν είναι εύκολη, αλλά μπορώ να σας πω ότι ακούσατε κύριε Βεσταγκέ πολλές επικοδομητικές ε, προτάσεις από τα μέλη της Επιτροπής καταλάβατε πολλές από τις ανησυχίες τους και των ψηφοφόρων τους. Με εντυπωσιάζει ότι ο κύριος Δέσ δέχτηκε πως οι Γάλλοι κάνουν καλύτερη δουλειά στην ε, αποσύνδεση των πληρωμών τους. Ε, είναι χώρο του κύριου Νταντέν βέβαια, αλλά πρέπει να σας πω ότι το 90% των πληρωμών της κοινής κοινωνικής πολιτικής είναι πλέον ε, αποσυνδεδεμένες στη Γαλλία. Μπορεί να κάνουν και κάποια εφελούσια κομμάτια αποδέσμευσης στις ορεινές περιοχές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό αλλά εν γέννη η μεταρρύθμιση ε, τουλάχιστον ως προς τους στόχους που ήθελαν οι νομοθέτες πηγαίνει σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν παραδείγματα στρέβλωσης ανταγωνισμών και γι' αυτό υπάρχουν οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Όταν υπάρχουν παραδείγματα στρέβλωσης του ανταγωνισμού πρέπει αυτές να εφαρμόνουν τους κανόνες. Κατά την άποψή μας έχουμε μια πολύ πιο ανταγωνιστική γεωργία παρότι έχουμε πολύ μεγαλύτερο επιπρόσθετο κόστος που συνδέεται με την βούλησή μας να έχουμε καλή ποιότητα τροφίμων, καλή ευημερία των ζώων, καλή προστασία του περιβάλλοντος. Προφανώς υπάρχει κόστος. Είναι ωστόσο ένα κόστος που κατά την άποψή μου είναι θετικό διότι παρουσιάζει την Ευρώπη σαν παραγωγό τροφίμων υψηλού, υψηλής ποιότητας που μπορεί να εξάγει σε τον κόσμο. Ξέρω ότι η συνάδελφος από το Εθνικό Μέτωπο διαφωνεί μαζί μου, αλλά δώσαμε στις περιφέρειες της Γαλλίας μεγάλη ευελιξία και σε όλες τις περιφέρειες δηλαδή για να μπορέσουν να παράσχουν επιπρόσθετη συνδεδεμένη υποστήριξη αν υπάρχει πρόβλημα με συγκεκριμένους γεωργούς. Αυτό είναι απόφαση κάθε κράτους μέλους να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που παρέχουν οι γεωργοί. Δεν δέχομαι λοιπόν ότι εγκαταλείψαμε τους μικρούς γεωργούς στην μεταρρυθμίση αυτή. Αυτό είναι τελείως λάθος, το απορρίπτω, δεν το δέχομαι. Επίσης θέλω να συμφωνήσω με κάποιους ομιλητές, τον κύριο Ντεκάστρο που μίλησαν για την ανάγκη να ε, υπάρχει μεγαλύτερος επαγγελματισμός των γεωργών για να μπορεί να συλλογικοποιηθούν τις διαπραγματεύσεις με την αλυσίδα φήμων αλλά και για τη διαθεσιμότητα τη χρήση των διαθέσιμων πόρων που η Ένωση παρέχει για τις οργανώσεις παραγωγών. Πρέπει σε πολλά κρατημέλη να προχωρήσουμε πολύ για να οδηγήσουμε στις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό έχει ιστορικούς λόγους. Θα προσπαθήσουμε την επόμενη διετία να πετύχουμε το στόχο της ε, καλύτερης ε, προώθησης στο εμπόριο, παρουσίασης των προϊόντων μας για να ανταγωνιστούμε με άλλους κλάδους, ιδίως οι μικροί γεωργοί. Συμφωνώ με αυτούς που ανέφεραν, το είπε και η κυρία για την ανάγκη να δούμε το θέμα του, τη, της παθητικής ίσπραξης των τιμών. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όχι μόνο την κυρία Βεστάγκερ αλλά και τον Βιερκόφσκι που είναι υπεύθυνο για τον αθέμητο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να συζητήσουμε με τον Επίτροπο για την διάσταση της γεωργίας στο πρόγραμμα εργασία του στο μέλλον. Προφανώς ε, δεν λειτουργεί το σύστημα όπως χρειάζεται. Είναι γεγονός ότι είναι δύσκολο να καταλάβουν πολλές φορές ε, κάποιοι ότι οι πρώτοι οι καταναλωτές γιατί η ζωή δεν βγαίνει σε νεκρό πέφτει η τιμή της πρώτης ύλη, αλλά δεν πέφτει το τελικό προϊόν. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που πρέπει να παρακολουθήσουμε, αλλά χρειάζονται στοιχεία για να κυνηγήσουμε κάποιου. Οι αρχέ ανταγωνισμού, κυρία Βεστάγκερ, θέλει στοιχεία. Αν υπάρχει ένα καρτέλ του Βόλου ε, ε, που ανέφερε ο κύριο Μακάρτη, πρέπει να έχουμε στοιχεία. Το είχαμε, είχαμε, είχαμε καταγγελίες στο παρελθόν, αλλά δεν είχαμε δεδομένα, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Άρα ευθύνη όλων μας είναι να παράσχουμε τα στοιχεία. Κάτι που δεν είναι εύκολο λόγω των, της μορφής των πρακτικών που ακολουθούνται. Κάνουμε κάτι για να εφαρμόσουμε αυτά που συμφωνήσατε. Ε, δεν ε, είναι σωστό να λέτε λοιπόν ε, ότι κάντε κάτι. Κάνουμε. Προσπαθούμε να εφαρμόσουμε αυτά που συμφωνήθηκαν στην πρόσφατη μεταρρύθμιση. Ωραίο είναι να μας λέτε κάντε κάτι. Τι. Εμείς κάνουμε. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με τη μεταρρύθμιση, αλλά εν τέλει δημοκρατική απόφαση είναι και αυτή την απόφαση εφαρμόζουμε. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Άγνου για την διστάμενη θέση που υπάρχει μεταξύ ασφάλειας τροφίμων αφενός και καταναλωτή αφετέρου. Χαμηλή τιμή δηλαδή που θέλει ο καταναλωτής. Πρέπει να, να εξισορροπήσουμε τις δύο αυτές αντί αντικρώμενες θέσεις. Το είπε πολύ σωστά ο ίδιος, λιγότερο σωστά εγώ. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουμε. Τι θα γίνει αν έρθει ας πούμε μας πλημμυρίσει η Βραζιλία με κάτι. Δεν το έχουμε προγραμματίσει αυτό ακόμα αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι ήδη έχουν πρόσβαση στην αγορά σε κάποιο μεγάλο βαθμό. Όχι όσο θα θέλανε αλλά έχουν πρόσβαση. Ίσως στο μέλλον να είχαμε, να θέλαμε, να θέλουμε να έχουμε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Βραζιλία γιατί έχουμε και επιθετικά συμφέροντα όχι μόνο άμυνα να πω και στον κύριο Φλάναγκαν ότι δεν, ε, δεν ερμηνεύει σωστά αυτό που είπα η αλεξάρτηση μεταξύ αστών κατοίκων της πόλης και κατοίκων της υπαίθρου δεν καλύπτεται σωστά από την κοινή γεωργική πολιτική αυτό το ξέρω αν δεν μιλήσουμε για βιωσιμότητα, υγιεινή ζωή, ηθική υποχρέωση παροχής διατροφής, ότι η τροφή δεν είναι μόνο γεωργία αλλά είναι βασικό κομμάτι της κοινωνίας, χάνουμε. Ο παραγωγός πρέπει να προσφέρει τρόφιμα όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχουμε υποχρέωση σαν ανταγωνιστική γεωργία να ανταποκρινόμαστε στη, στα αιτήματα του αυξανόμενου πληθυσμού ανά τον κόσμο πρέπει να θρέψουμε. Αυτή την υποχρεώση πρέπει να την καταλάβουν και οι πολίτες και οι κάτοικοι των πόλεων και οι κάτοικοι της υπαίθρου. Κλείνω ευχαριστώντας τα μέλη για τη συνεισφορά τους. Δεν, δεν απάντησα σε όλους ατομικά, πήρα σημειώσεις πάντως και θα απαντήσουμε στο τελικό κείμενο που θα βγει τον Οκτώβριο, το φθινόπωρο, συγγνώμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Η κυρία Πίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι μεγάλωσα 300 μέτρα μακριά από τον πρώτο συνεταιρισμό γαλακτοκομικών του κόσμου. Και ο λόγος που συνεταιρίστηκαν τότε οι αγρότες ήταν γιατί ήθελαν να είναι πιο επαγγελματίες, να επενδύσουν περισσότερα και να πάρουν καλύτερες τιμές για τα προϊόντα τους. Είναι μια πολύ απλή και βασική συλλογιστική που λειτουργήσε τότε και θα λειτουργήσει και τώρα. Και θεωρώ ότι είναι ένα πολύ ισχυρό ε, μήνυμα ε, το σημερινό, ότι δηλαδή θα αξιοποιήσουμε αυτές τις κατευθυντηρίες γραμμές για να πετύχουμε αυτόν τον στόχο, να μπορούν να συνεταιρίζονται, να συνοργανώνονται ε, μαζί οι παραγωγοί να βάζουν, να συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους αλλά να μην πάνε σε κρυφά μονοπωλιακά παιχνίδια. Και ελπίζω ότι θα επανέλθουμε για να δούμε κατά πόσο λειτουργεί αυτό το πράγμα, γιατί είναι κοινή μας αρμοδιότητα ως συνομοθέτες. Σας ευχαριστώ για τη συνεδρίαση με ενέπνευσε ήδη και ε, σας παρακαλώ να μας αναγκάσετε να εμείνουμε στην υπόσχεση που σας δώσαμε ότι δηλαδή θα εκδώσουμε κατευθυντήριες γραμμές που να είναι ε, χρήσιμες και να μπορούν να αξιοποιηθούν. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Ας αξιοποιήσουμε αυτή την πρόταση της ε, αξιότιμης ε, κυρίας Επιτρόπου για να διαβιβάσουμε γραπτός ε, τις διάφορες παρατηρήσεις και τα σχόλια των μελών της κοινοβουλευτικής μας επιτροπής. Αυτό θα μας βοηθήσει όλους. Μπορούμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να εκφράσουμε τη γνώμη μας πιο συγκεκριμένα. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο σε αυτή την ε, συνεδρίαση της μιάμισης ώρας για το θέμα αυτό. Μπορούμε λοιπόν να συμβάλλουμε στη συζήτηση γραπτός και χαίρομαι διότι βλέπω ότι και άλλοι επίτροποι ασχολούνται με το θέμα της γεωργίας εκτός από τον δικό μας επίτροπο. Αυτό είναι πολύ καλό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερο και το επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά για την παρουσία της αξιότιμης κυρίας Επιτρόπου εδώ στην Επιτροπή μας. Της Επιτρόπου που έχει το χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού, το εξαιρετικά σημαντικό χαρτοφυλάκιο του ανταγωνισμού και θα σας ξανακαλέσουμε και θα καλέσουμε και άλλους επιτρόπους στην Επιτροπή εδώ την Κοινοβουλευτική διότι πρέπει να διευρύνουμε τις γνώσεις μας και να εξετάσουμε την αγορά της γεωργίας υπό όλες τις δυνατές πτυχές. Ο κύριος Κάστρο μίλησε για την πολύ ασθενή δύναμη των αγροτών. Έχουμε πολλά παραδείγματα που δείχνουν πόσο διαφορετικές είναι οι τιμές που παίρνουν οι αγρότες από τη μία και οι τιμές τις οποίες διατίθεται τα προϊόντα στους καταναλωτές από την άλλη. Σε μερικές περιπτώσεις η απόκληση είναι τεράστια. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους δύο επιτρόπους. Με τον κύριο Χόγκαν τα λέμε σχεδόν καθημερινώς. Αλλά κυρία Φρεστάγκερ θα σας καλέσουμε του χρόνου ίσως σε δύο χρόνια, δεν ξέρω, για να κάνουμε έναν απολογισμό όλες αυτές τις συνεργασίες και τις δράσεις. Προτείνω δύο-τρία λεπτά διακοπή για να οργανωθούμε για την ψηφοφορία. Ο εισηγητής ε, ήδη έχει έρθει, ο κύριος Νίκολσον. Ευχαριστώ τους δύο επιτρόπους και τρία λεπτά διακοπή πριν συνεχίσουμε παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, καθίστε, θα ξεκινήσουμε την εξέταση του δεύτερου σημείου της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για τη ψήφιση της έκθεσης του κυρίου Νίκολσον για το μέλλον του γαλακτοκομικού τομέα στην Ευρώπη, απολογισμός της υλοποίησης της δέσμης μέτρων για το γάλα. Κυρίες και κύριοι, Ίσως ε, είναι καλό να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Νίκολσον, ο οποίος θα μας κάνει την παρουσίαση αυτού του θέματος. Παρακαλώ. Κύριε Νίκολσον, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε ότι ούτε δύο λεπτά δεν θα κάνω. Έχω ιστορικό ταχύτητος και συντομίας. Να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους εισηγητές, στους και όλες εισηγητές με συγχωρείτε, στη γραμματεία, σε όλους όσοι με βοήθησαν σε αυτή τη διαδικασία. Τους ευχαριστώ για τόσες τροπολογίες που καταφέραμε να ε, ε, δημιουργήσουμε συμβιβαστικές ε, τροπολογίες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Βεβαίως δεν υπάρχει σύγκληση 100%. Να ευχαριστήσω το προσωπικό του γραφείου μου και της πολιτικής μου ομάδας για τη βοήθεια που μου παρήχαν. Όλοι γνωρίζουμε ότι είναι πλέον αργά, Δευτέρα βράδυ. Δεν θέλετε από μένα ε, μακροσκελής ομιλίες. Ωστόσο, δύο δευτερόλεπτα αξίζει να μοιραστώ μαζί σας το εξής. Το 89 που έγινα μέλος αυτής της Επιτροπής, η Ευρώπη είχε βουνά γάλακτος και άλλων προϊόντων να σαπίζουν. Όλα αυτά δεν υπάρχουν πια. Είναι διαφορετική αγορά και πρέπει να ε, προσαρμοστούμε, πρέπει να είμαστε ηγέτες παγκοσμίω και όχι να ακολουθούμε τις παγκόσμιες εξελίξεις. Πρέπει εμείς να ηγηθούμε. Να ευχαριστήσω ξανά όλους και όλες. Έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά, να αφήσουμε το σήμα μας, το χαρακτηριστικό μας γνώρισμα και ελπίζω να συμφωνήσετε και να υπερψηφίσετε την έκθεσή μου. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Πράγματι. Πολύ ωραία η ευχή σας. Να έχουμε τη φιλοδοξία να ηγηθούμε σε αυτές τις εξελίξεις παγκοσμίω. Κυρίες και κύριοι, εάν υπάρχει προφανής πλειοψηφία, δεν θα ζητώ να μου πείτε ποιος είναι κατά και ποιος απέχει. Αλλά βεβαίως μπορείτε να παρεύετε, δεν θέλω να αλλάξω καθόλου τη βούλησή σας όταν ψηφίζετε. Το λέω για να είμαστε πιο γρήγοροι και πιο αποτελεσματικοί. Υπάρχουν πολλές συμβιβαστικέ τροπολογίες και οι εκπρόσωποι των διαφορετικών πολιτικών ομάδων έχουν, συμμετάσχει στις συζητήσεις για αυτές τις συμβιβαστικέ τροπολογίες. Δεν υπήρξε συμφωνία 100% αλλά έτσι είναι η δημοκρατία. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά τις συμβιβαστικέ τροπολογίες ή για ανατάσεως χειρός. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ. Ε, ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία της Επιτροπής Ελέγχου Μπέκερ. Ποιος είναι υπέρ κατά απορρίπτεται. Τροπολογία της ε, Κοκομπού, Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Το σί υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Η τροπολογία 2, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τρία, Τροπολογία Ριμπέιρο υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Η τέσσερα, υπέρ, ευχαριστώ, εγκρίνεται. Η πέντε, υπέρ, την πέντε. Θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Ε, ξεκινάει η ψηφοφορία για την ε, ε τροπολογία πέρας για την τέσσερα εγκρίνεται. 5. Ποιος είναι υπέρ της 5. Κατά. Απορρίπτεται. 6. Υπέρ. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 9. Υπέρ Κατά. Απορρίπτεται. 10 και 11. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ εγκρίνεται. 12 υπέρ. Εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία α1. Ποιος είναι υπέρ. Δια της ηλεκτρονικής οδού άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 82. Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 83 υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 94α. Όχι, 94. Συμβιβαστική τροπολογία α2. Με συγχωρείτε. Συμβιβαστική τροπολογία α2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Πάμε στην 94. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 95 υπέρ, Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α3. Άρχεται η ψηφοφορία για της ηλεκτρονικής οδού. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Πάμε στην 108. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι κατά. Απορρίπτεται. 109 υπέρ. Εγκρίνεται. 112 υπέρ. Κατά. επαληθεύουμε δια της ηλεκτρονικής οδού. Άρχεται η ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α4. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 122. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Πάμε. 162. Ποιος είναι υπέρ. Όχι, θα την επαληθεύσουμε για τη ηλεκτρονική οδού άρχεται η ψηφοφορία για την 162. Πέρα της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 162. Πάμε στη, στη συμβιβαστική τροπολογία Α5. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 136. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Πάμε στη συμβαστική Α6. Όχι, συγγνώμη, λέει ο Πρόεδρος. Συμβιβαστική τροπολογία Α5 μικρό α. Ε, ξεκινάει ηλεκτρονική ψηφοφορία για το 5α μικρό. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε συμβαστική ε, α6. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας της ε, ψηφοφορίας εγκρίνεται. 427. Ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 146 τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 148 υπέρ. Εγκρίνεται. 149 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 152 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6α μικρό. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστώ. 304. Ποιος είναι υπέρ της 304. Εγκρίνεται. 401. Υπέρ κατά απορρίπτεται 402 υπέρ κατά εγκρίνεται 443 ε, υπέρ εγκρίνεται 153 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική α7 Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 164. 164. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 156 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά απορρίπτεται 168 αποσύρεται 169 υπέρ κατά απορρίπτεται 170 υπέρ εγκρίνεται 172 υπέρ εγκρίνεται 173 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Ευχαριστώ. Συμβιβαστική 9α. Ε, άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Ευχαριστώ εγκρίνεται. Πάμε στην 187 υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 190 υπέρ. Εγκρίνεται. 191 κατά. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά απορρίπτεται. 197 υπέρ, εγκρίνεται. 200 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, ε, τροπολογία υπαριθμών 10. Ε, η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 206 υπέρ. Κατά. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικός. Ξεκινά η ηλεκτρονική ψηφοφορία για την 206. Του κυρίου Ταραμπέλα. Πέρος, πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 25 κατά. 25 ψήφοι κατά. 207 υπέρ εγκρίνεται 202 υπέρ εγκρίνεται 210 υπέρ 211 υπέρ κατά απορρίπτεται Τροπολογία της Επιτροπής για τον έλεγχο του προπολογισμού συμβαστική Ποιο είναι υπέρ η 6 εγκρίνεται ε, η 7 της Ιδίας Επιτροπής υπέρ κατά εγκρίνεται 8 υπέρ κατά απορρίπτεται 9 υπέρ κατά δεκτή 10 υπέρ κατά απορρίπτεται 212 υπέρ δεκτή συμβιβαστική α11 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 220 τοπολογία υπέρ κατά απορρίπτεται 221, 222, 223 υπέρ. Ευχαριστώ κατά. Απορρίπτεται. Απορρίπτονται και οι τρεις. 224 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 225 υπέρ. Εγκρίνεται. 226 Διορθώνει ο πρόεδρος. ...246 τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Απολύπτεται. 227 υπέρ. Κατά. Δεκτή. Συμβιβαστική α12 Άρχεται η ψηφοφορία. τη ψηφοφορία. Δεκτή. 244 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 247 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική α13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 260 τροπολογία. Υπέρ. 260 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 261 υπέρ. Δεκτή. 265 υπέρ κατά απορρίπτεται 266 υπέρ δεκτή 267 υπέρ κατά απορρίπτεται 268 υπέρ κατά απορρίπτεται διορθώνει ο πρόεδρος ηλεκτρονικός έλεγχος για την 268 Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 270 υπέρ. Δεκτή. 262 υπέρ. Δεκτή. 272 υπέρ. Δεκτή. Τώρα, η 275 υπέρ, 275 υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 276 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α15. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρα ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτεί. 298 τροπολογία υπέρ. Κατά. Συγγνώμη, ε, πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος 298 άρχεται η ψηφοφορία για το 298 εγκρίνεται συμβιβαστική α17 άρχεται η ψηφοφορία Μιλάω γρήγορα φαίνεται που μπλοκάρει την ψηφοφορία. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να μιλήσω πιο αργά. Λοιπόν, συμβιβαστική α17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. 305 τροπολογία υπέρ. Ευχαριστώ. Εγκρίνεται. 308 υπέρ. Δεκτή. 309 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 311 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 312 υπέρ. Δεκτή. 313 υπέρ κατά απορρίπτεται 314 υπέρ κατά απορρίπτεται 315 υπέρ κατά απορρίπτεται 316 υπέρ κατά απορρίπτεται 317 υπέρ κατά απορρίπτεται 318 υπέρ κατά απορρίπτεται. Συμβιβαστική α18 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 331 υπέρ κατά απορρίπτεται. 332 υπέρ κατά απορρίπτεται. 333 υπέρ κατά απορρίπτεται 334 υπέρ κατά απορρίπτεται 335 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική α19 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Τροπολογία τώρα 344. Υπέρ. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Α20. Άρχεται ψηφοφορία. Θα γίνει έλεγχος πρώτα για την 344 ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. βιβαστικη Συμβιβαστική Α20 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 372 τροπολογία υπέρ κατά απορρίπτεται 373 τροπολογία υπέρ κατά απορρίπτεται 374 υπέρ κατά απορρίπτεται 375 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίφθηκε θα κάνουμε έλεγχο για την 375 ηλεκτρονικό έλεγχο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Με τρει ψήφου διαφορά. 376 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 377 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Α21. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ευχαριστώ, εγκριθήκε. Συμβιβαστική Α22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ε, ευχαριστώ, εγκρίνεται. Τροπολογία 389 υπέρ δεκτή. Τροπολογία 390 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 271 υπέρ, εγκρίνεται. 382 υπέρ, δεκτή. 403 συγγνώμη υπέρ, Ε, α23. Συμβιβαστική α23. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 403 δεν ψηφίζουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε η συμβιβαστική α23. Τροπολογία 396. Υπέρ. Δεκτή. 393 δεύτερο τμήμα υπέρ Δεκτό. Η 404 αποσύφηκε. 405 υπέρ. Δεκτή. 406 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 407 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 408 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 409 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική α24 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ευχαριστώ 425 υπέρ ευχαριστώ δεν κρίνεται 426 υπέρ κατά απορρίπτεται 428 υπέρ κατά απορρίπτεται 429 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική α25 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται απολογία <clears throat> 439 Τρίτο τμήμα. Υπέρ. Δεκτό. 441 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 442 υπέρ. Δεκτό. 444 υπέρ. Δεκτή. Α26. Συμβιβαστική. Δεκτή. 447 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίφθηκε θα γίνει έλεγχος όμως πέρας ψηφοφορίας 448 υπέρ δεκτή 458 συγγνώμη συμβαστική α27 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας ευχαριστώ η 473 υπέρ κατά απορρίπτεται 476 Υπέρκατα κατά θα γίνει έλεγχος για την 476 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας δεκτή 471 κατά υπέρ κατά απορρίπτεται 478 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 468 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 469 υπέρ, έλεγχος για την 468 ηλεκτρονικά, άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται η 468. 4.82 82 το υπολογία τώρα. Υπέρ. Δεκτή, ευχαριστώ. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβιβαστική R1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 22. Υπέρ, Ευχαριστώ. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική ερώ 2. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέραση οφορία Εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά απορρίπτεται 39 υπέρ κατά απορρίπτεται 40 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβιβαστική R3 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας δεκτή 44 τροπολογία 46 διοθώνει ο πρόεδρος. Διοθώνει ξανά ο πρόεδρος. 44. Υπέρ του 44. Κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 45. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 46. Υπέρ κατά απορρίπτεται. 47. Υπέρ δεκτή. 48 καταπίπτει. σαραντοκτω υπέρ. Ευχαριστώ δεκτή. 49 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 51, ταραμπέλα. Υπέρ, κατά, δεκτή. Συμβαστική R5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Δεκτή. Τροπολογία 53, υπέρ. Δεκτή. Πενήντα υπέρ δεκτή 60 υπέρ κατά απορρίπτεται 61 υπέρ κατά απορρίπτεται 62 υπέρ κατά απορρίπτεται 75 υπέρ κατά απορρίπτεται 63 υπέρ κατά Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Ρο 6. Ήθελα να ζητήσω η τροπολογία 70 να ψηφιστεί χωριστά. Δεν είναι κομμάτι του συμβιβασμού. Ψηφίζουμε για το R6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η συμβαστική πρόταση. Στην τοπολογία 70 της κυρίας Μόη. Υπέρ κατά θα γίνει έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία για την 70 πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 71 υπέρ δεκτή. 72 υπέρ εγκρίνεται. 73 υπέρ Εβδομήντα τέσσερα υπέρ κατά καταπίπτει το τροπολογία αυτή λέει ο πρόεδρος 76 υπέρ κα, απορρίπτεται 77 υπέρ κατά για την 77 ψηφίζουμε άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά για την 77 πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 78 απορρίπτεται σχέδιο ψηφίσματος ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται να ευχαριστήσω τους ε, συμμετέχοντες ε, στην πολύ αποτελεσματική αυτή διαδικασία ψηφοφορίας και να συγχαρώ τον εισηγητή. Κύριε Νίκολσον, θέλετε να πείτε δύο λόγια. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, νομίζω ότι πολύ αποτελεσματικά ολοκληρώσαμε τις ψηφοφορίες, αλλά θα ήθελα να πω το εξή, ότι νομίζω ότι όλοι στην αίθουσα γνωρίζουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο γαλακτοκομικός τομέας στο σύνολο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και θα ήθελα όχι να έχουμε μόνο διμερή διάλογο, αλλά να έχουμε πλήρη συζήτηση στην Ολομέλεια και να επιτρέψουμε στα μέλη της Επιτροπής μας να εκφράσουν τη γνώμη τους όχι μόνο πάνω στην έκθεση αυτή αλλά και σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τομέας ε, του γάλακτος σε όλη την Ευρώπη. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ λοιπόν ε, να προωθήσετε το θέμα αυτό και θα παρακαλούσα και τους επικεφαλείς των ομάδων στη διάσκεψη των ΟΕΔΡων ε, να φροντίσουν να έχουμε πλήρη συζήτηση για το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ όλους για την υπομονή και επιμονή σας. Νομίζω ότι το ολοκληρώσαμε πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικό από ό,τι νομίζαμε. Σα ευχαριστώ όλου για τη συμμετοχή. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή. Κυρίες και κύριοι, ήταν μακρά η συζήτηση. Όλοι πρέπει να είναι δραστήριοι στη δική τους πολιτική ομάδα γιατί όλοι πρέπει να έχουν συνείδηση της σημασία των προβλημάτων του γαλακτοκομικού τομέα. Αυτό πρέπει ε, να αντιμετωπίσουμε ως πρόκληση. Εμείς το γνωρίζουμε αλλά θα πρέπει να το μάθουν κι άλλοι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, ψηφοφορία. Ζητώ συγγνώμη για το γεγονό ότι συνεδριάσαμε τόσο αργά το βράδυ αλλά ήταν η μόνη δυνατότητα. Ευχαριστώ τον εισηγητή, τους συμμετέχοντες, τους σκιώδεις εισηγητές και τους διερμηνείς. Ευχαριστώ.